Euh, Επαναλαμβάνονται οι εργασίε της Επιτροπής. Για όσους δεν ήταν το πρωί εδώ να τους καλημερίσω, να χαιρετήσω τα μέλη του συνεδρίου που ήρθαν, τον Γενικό Διευθυντή του Υπηρεσία Καταπολέμησης των Απατών, θα του δώσω αμέσω το λόγο και θα μιλήσουμε για το σημείο 7. Αλλά πριν να μιλήσουμε γι' αυτό, να σας πω ότι ο πρόεδρο μα έρχεται από τι κάτω χώρε και θα πρέπει να έρθει μέσα στο απόγευμα αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα. Ε, ανάμεσα στις 4 ε, και το τέλος της συνεδρίασης. Σημείο 7 λοιπόν. Έκθεση 2011 του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας της Απάτης και δίνω τον λόγο στον κύριο Κέσλερ, Γενικό Διευθυντή της εν λόγω υπηρεσίας. Σας ευχαριστώ. Δύο λόγια και μετά φαντάζομαι. Ελπίζω ότι θα έχετε ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Πρώτη μου παρουσίαση ετήσιας ε, έκθεσης ε, για τις δραστηριότητές μας, αλλά όπως ξέρετε η, πρόκειται, η έκθεση αυτή αφορά τις δραστηριότητες του 2010 της Όλαφ. όταν δεν ήμουν ακόμα επικεφαλή δηλαδή της υπηρεσίας. Παρουσιάζω λοιπόν το έργο το προκατόχου μου. Αλλά νομίζω πως μπορούμε να βρούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και νούμερα, κάποια θέματα τα οποία θα είναι ενδιαφέροντα σε σχέση με την παρούσα διαδικασία μεταρρυ... νομοθετικής μεταρρύθμισης καθώς και ενδιαφέροντα ζητήματα και διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε για τον εσωτερική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας την οποία αυτή τη στιγμή κάνουμε. Πρώτο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας όσον αφορά τις έρευνες. Αν δείτε, έχουμε περίπου χιλιάδες εισερχο... ε, χίλιες εισερχόμενες πληροφορίες ετησίως. Το ίδιο συνέβη και το 2010 και από αυτές τις χίλιες υποθέσεις που ανοίξαμε ξεκίνησαν 150 έρευνες συν 75 υποθέσεις συντονισμού και βοήθειας. Αυτό το νούμερο είναι πάνω κάτω λογικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω πως κάτι λέει. Ότι δηλαδή πάνω κάτω μόνο 20% των εισερχόμενων πληροφοριών έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον λιγότερο από το 25% των ε, πληροφοριών που λαμβάνουμε οδηγούν σε έναρξη έρευνας. Στο μέλλον λοιπόν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση, να αυξήσουμε δηλαδή την ποιότητα των εισερχόμενων πληροφοριών. οι ανοιχτέ γραμμές για το κοινό που μπορεί να καλέσει και να δώσει πληροφορίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να καταστήσουν δυνατό τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο να καταστήσουν δυνατή τη χρήση της Όλαφ και την ενημέρωση της Όλαφ εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση για απάτη ή για διαφθορά. που ζημιώνει το ευρωπαϊκό συμφέρον. Μόνο 46% των εισερχόμενων πληροφοριών, από αυτές τις χίλιες εισερχόμενες πληροφορίες, μόνο το 46% προέρχεται από τον δημόσιο τομέα, δηλαδή ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εθνικές αρχές. Και αν εξετάσουμε προσεκτικά τα εθνικά στοιχεία για ορισμένα κράτη-βέλη, μάλιστα δεν έχουμε καμία πληροφορία. Πράγμα το οποίο δεν είναι και πολύ πιστευτό, γιατί είναι μάλλον απίθανο σε κάποια κράτη να μην υπάρχει ούτε μία περίπτωση, ούτε μία υπόθεση που να ενδιαφέρει την Όλαφ. Συμφωνείτε κυρία Γκρέσλε, ναι. I must say that Έλεγα λοιπόν ότι κανονικά δεν έχουμε αυτόν τον αριθμό στην έκθεση, αλλά μπορώ να σας το πω προφορικά ότι η ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τον δημόσιο τομέα είναι πολύ ψηλότερη από την μέση ποιότητα πληροφοριών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε Ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες χρειάστηκε να ενθαρρύνω τις εθνικές αρχές αρχές αρμόδιες ε, για, την, ε, για τις δαπάνες αλλά και τις ε, εθνικές αρχές επιβολής της τάξης να αναφέρονται στην όλα όταν έχουν πληροφορίες για απάτη που μπορεί να μην εξεταστούν απόλυτα σε εθνικό επίπεδο. Και για να δώσουμε κάποια κίνητρα σε αυτές τις υπηρεσίες, μπορώ να σας πω ότι στην επόμενη έκθεση θα έχουμε πιο ξεκάθαρα στοιχεία ανά κράτος για το πόσες πληροφορίες προέρχονται αναχώρα, πόσες πληροφορίες αναχώρα έρχονται από το δημόσιο τομέα και πόσες από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το νούμερο θα είναι ενδιαφέρον για να δούμε ποιος βαθμός συνεργασίας υπάρχει από το κάθε κράτος μέλος. Γιατί αν για κάποιο κράτος μέλος έχει ένα σωρό πληροφορίες για απάτες, αλλά από τον ιδιωτικό τομέα και όχι από τον δημόσιο τομέα, αυτό σημαίνει πως η χώρα αυτή έχει πρόβλημα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. We move to another point we of our cases, of our investigations, actually. Uh, Το σύνολο της διάρκειας μιας υπόθεσης από τότε που φτάνει η πληροφορία μέχρι την εκπόνηση της τελικής έκθεσης περί της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι 27,9 μήνες. Αν με ρωτήσετε τι σημαίνει κόμμα 9, δεν ξέρω ακριβώς σημαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για πάνω από 27 μήνες διάρκεια. Speaking, I don't know, nine days or... Oh, okay. Ah, okay, okay, okay. So actually it's almost uh, so it's 27 months. Είναι 27 μήνες και 27 μέρες δηλαδή. Δηλαδή αυτή είναι η μέση διάρκεια διερεύνησης μιας υπόθεσης. Δεν είναι και πολύ ωραίο νούμερο. Αλλά ξέρετε ήδη ότι η μέση διάρκεια ε, διερεύνησης μιας υπόθεσης είναι αρκετά μακριά. Πρόκειται ωστόσο για μια νομοθεσία που ισχύει εδώ και πέντε χρόνια. Παλιότερα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Βελτιωνόμαστε, αλλά όχι αρκετά. Πιστεύω λοιπόν, και το λέω ενώπιόν σας, θα μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, πως 27, καν 28 μήνες είναι πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Βέβαια, οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται κάπως στην Όλαφ, αλλά όχι απόλυτα στην Όλαφ. Ένας από τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η μεγάλη διάρκεια οφείλεται στους εταίρους μας. Δηλαδή τα κρατημέλη, τα οποία ιδιαίτερα κατά την αρχική φάση της αξιολόγησης καθυστερούν να απαντήσουν, οι εθνικές αρχές δηλαδή καθυστερούν να απαντήσουν οι αρχές αρμόδιες περί των δαπανών όταν τους ζητάμε πληροφορίες για την ε, δαπάνη ευρωπαϊκών χρημάτων. Τι βασικές πληροφορίες δηλαδή που χρειαζόμαστε για να αποφασίσουμε αν θα αρχίσουμε ή όχι έρευνα. Επίσης μας παίρνει χρόνο το να διακρίνουμε ποιες πληροφορίες είναι χρήσιμες ή όχι για να ξεκινήσουμε μια διερεύνηση. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως αυτό παίρνει και ένα χρόνο μέχρι που να πάρουμε τις αρχικές βασικές πληροφορίες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Ίσως η της υπηρεσίας βασικά έχει να κάνει με αυτό το νούμερο και με το στόχο της μείωσης της διάρκειας ε, διεκπαιρέωσης μιας ε, υπόθεσης. Καταρχήν εμείς ε, θα είμαστε πιο ενεργοί απέναντι στα κράτη-μέλη ε, ώστε να παίρνουμε τις πληροφορίες πιο γρήγορα. Δεν θα στέλνουμε απλά μια επιστολή και μετά θα περιμένουμε για μια άλλη επιστολή. Θα τους ζητάμε να πρόσβαση στα βάση δεδομένων. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο ένα θέμα πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων. Ήδη έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα παρόμοιο θέμα, αλλά αυτές είναι βάσεις δεδομένων που σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι ανοιχτέ. Θα πρέπει να είναι ανοιχτέ. Και είναι οι βάσεις δεδομένων που αφορούν την χρηματοδότηση από την Ένωση. Τα ευρωπαϊκά χρήματα δηλαδή που δαπανώνται σε εθνικό επίπεδο. Και έτσι να μπορούμε να είμαστε πιο γρήγοροι για να διακρίνουμε από τις εισερχόμενες πληροφορίες σε μερικές εβδομάδες, αντί για μήνες ή και χρόνια. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε ένα διαφορετικό οργανόγραμμα για την Όλαφ Δημιουργούμε μια νέα μονάδα, που θα, ένα νέο τμήμα που θα ασχολείται μόνο με τη φάση της αξιολόγησης, δηλαδή τη φάση επιλογής αποκλειστικά. Έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μειώσουμε αυτή την περίοδο που τώρα υποτίθεται ότι διαρκεί 4 μήνες, ενώ κατά μέσο όρο διαρκεί 8. Θα έχουμε λοιπόν αυτή την ε, νέα μονάδα, η οποία επίσης θα δώσει συνοχή στη διαχείριση των εισερχόμενων πληροφοριών. Σήμερα οι εισερχόμενες πληροφορίες αντιμετωπίζονται σε αρχικό στάδιο σε μια εκπεριτροπήση, μαλλον τυχαια βαση απο διαφορες ερευνητικες μοναδες στο μελλον η το ερευνητικό τμήμα αυτό θα ασχολείται μόνο με την διαδικασία αυτή επιλογής και έτσι θα προβαίνουμε ταχύτερα στη φάση της ε, πραγματικής έρευνας. Εν πάση περιπτώσει είναι μια διοικητική επόφαση ώστε σε ένα ή μάλλον σε δύο χρόνια θα δούμε κατά πόσο η ιδέα αυτή ήταν επιτυχής, όπως ελπίζω, ώστε να συντομευθεί αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελευταία παρατήρηση, τελευταίο στοιχείο, επί το οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, είναι τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Όλαφ αν θέλουμε να δούμε όχι τα πλήρη, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια σημαντικά αριθμητικά στοιχεία, που είναι τα αποτελέσματα από δικαστικής άποψης, αλλά και από οικονομικής άποψης. Δικαστικά, uh, Δικαστικά αποτελέσματα να σας πω ότι ως αποτέλεσμα των ε, ρευνών της Όλαφ το 2010 συνολικά απαγγέλθηκαν ποινές που ανέρχονται σε σύνολο 125 ετών φυλάκιστης και η, τα πρόστιμα είναι 1,5 δις που επιβλήθηκαν. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακτήσει ε, σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα των ερευνών. Να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτά τα νούμερα που περιέχονται στην έκθεση του 2010 ως αποτέλεσμα των ερευνών της ΟΛΑΦ ε, ε, αφορούν ε, τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών γιατί κανονικά περνάνε κάποια χρόνια μέχρι σότου μάλλον ανάμεσα στην έκδοση της έκθεσης της ΟΛΑΦ που αποστέλλεται στο Εθνικό Δικαστικό Σώμα ή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ανάκτηση των χρημάτων. ή στην κατάληξη σε μια εθνική απόφαση από εθνικό δικαστήριο. Αυτά τα νούμερα λοιπόν δεν λένε και πολλά πράγματα για τις δραστηριότητες του 2010 αυτού καθ' αυτού. Καταγράφηκαν το 2010, αλλά πρόκειται για έρευνας που έκανε η όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσω ότι είναι πολύ καλά αποτελέσματα δεν είναι τα μόνα αποτελέσματα, δεν είναι τα πλήρη αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Όλαφ γιατί πιστεύω και ελπίζω πως οι δραστηριότητες της Όλαφ έχουν και ένα ε, αποτρεπτικό χαρακτήρα, προληπτικό Ε, απέναντι στους απατεώνες και γενικότερα στο προσωπικό της Ένωσης, δίνοντας τα καλά παραδείγματα, αποτρεπτική, αποτρεπτικό δηλαδή αποτέλεσμα επιρροή που δεν μπορεί να μετρηθεί. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μετρήσιμα στοιχεία για τη δραστηριότητά μας. Που, κατά τη γνώμη μου, δείχνουν πως η Όλαφ είναι απαραίτητη και τα χρήματα που δαπανώνται από την Όλαφ ε, δαπανώνται Σωστά, γιατί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ανακτούν περισσότερα χρήματα από όσα κοστίζει η λειτουργία της Όλαφ. Αυτά λοιπόν και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Merci, euh, Σας, ευχαριστώ. κύριε Γενικά Διευθυντά. Θα προτείνω να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, στον κύριο Βαλσέτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Μας παρουσιάσατε την έκθεση με λεπτομέρεια. Μας παρουσιάσατε και κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία εκ πρώτης όψεως μας φαίνονται πολύ καλά. Θα πρέπει να σας συγχαρώ για τα καλά σας αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι εσείς αναλάβατε καθήκοντα σας το 2011, από ό,τι είπατε. Ένα από τα βασικά θέματα, θεωρώ, είναι το εξή. Ο αριθμός των ε, υποθέσεων έρευνας έχει μειωθεί και η περίοδη διεξαγωγή τη έρευνα έχουν μειωθεί. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσει. Γιατί ένα από τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, παρά τα, αριθμητικά στοιχεία, είναι το εξή. Μέχρι το 2010, η Όλαφ αποφάσισε, κατέληξε σε ένα ποσό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά σε ποσό ανάκτησης έχουμε φτάσει μόνο το 1 δις. Είσαστε το θεσμικό όργανο που διεξάγει τέτοιες έρευνες και ασφαλώς συνεργάζεστε με τα κράτη-μέλη, με τις δικαστικές αρχές και αναφέρατε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στη συνεργασία αυτή. Και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα από τα προβλήματα για το ότι τα κράτη-μέλη δεν ανοίγουν, αν θέλετε, τα... δεν δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία τους. Αλλά μόλις σας δοθεί τέτοια πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, θα έχετε πιο μεγάλο όγκο εργασίας. Κάποιες ερωτήσεις έχω σημειώσει. Οι οποίες όμως είναι ίσονος σημασίας. Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων, η συνεργασία μεταξύ των διάφορων θεσμικών οργάνων, γύρω τζάστ και γύρω για παράδειγμα και άλλη μια πτυχή είναι η στάση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητές σας, τις εργασίες σας. Ασφαλώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται συνεργασία και το πρωί άλλωστε κάναμε μια συζήτηση για την ανεξαρτησία της Όλαφ. Όλοι είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συμφωνία για κάποιες βασικές αρχές, για κάποιους βασικούς κανόνες και αυτό ενδεχομένως να διευκολύνει το έργο σας και να το κάνει και πιο εύκολα κατανοητό στον κόσμο. Σήμερα λοιπόν θεωρώ ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι το εξή. κρατεμέλη παρουσιάζουν πολλές ε, ατασταλίες, κρατημέλη, συγκεκριμένα η Ρουμανία, η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Πολωνία παρουσιάζουν 60% να πληροφορίες που έχουν να κάνουν με ατασταλίες. Αναρωτιέμαι, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν λανθασμένες πρακτικές στις χώρες αυτές ή μήπως έχουν τεθεί λάθος ερωτήσεις ή μήπως έχουν τεθεί ερωτήσεις με λάθος τρόπο. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, η Βουλγαρία και ο τομέας ο γεωργικός έχουν διεξαχθεί 81 έρευνες. Και 61 εξ αυτών έχουν να κάνουν με τον γεωργικό τομέα. Ενώ στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια ήταν διαφορετικό το ποσοστό αυτό. Ήταν μόνο 26 οι περιπτώσεις αυτές στο σύνολο των υποθέσεων. Στο μέλλον θα συζητάσουμε πιο πολύ θέματα ε, επιδοτήσεων και γεωργίας και θεωρώ ότι είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες. Ύστερα, ε, χώρες όπως το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Έχουν υπάρξει μειώσεις της τάξης του 50% τα τελευταία χρόνια. Γιατί? Κάτι άλλο το 2010 για τις άμεσες ε, εργασίες σας αφιερώσατε 37% του χρόνου εργασίες σας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα σωστό ποσοστό. Αυτό σκοπεύετε να κάνετε και στο μέλλον και θεωρείτε ότι ο χρόνος που δαπανήθηκε για έρευνα ήταν επαρκής. Αυτά ήταν τα βασικά ερωτήματα που ήθελα να σας θέσω. Ανυπομονώ να ακούσω τις απαντήσεις σας και ανυπομονούμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε για το 2011. Νομίζω ότι θα σημειωθούν καλά αποτελέσματα και σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Καδιευθυντά Κιάσλα, αναφερθήκατε σε εννέα προκλήσεις ε, και σε καινούριε προκλήσει επίση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Όλαφ και ε, για τι οποίε ε, δεν θα αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται. Ξέρουμε εμεί που ασχολούμαστε με τον προπολογισμό ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά. Γι' αυτό ρωτώ. Ποιε είναι οι καινούριε πρωτοβουλίε που προβλέπετε στην Όλαφ. Έχετε σκεφτεί καθόλου πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι και πώς θα ανακατανεμηθούν στον, στην υπηρεσία σας. Κύριε Γενική Διευθυντά, ευχαριστώ. Τα κράτη-μέλη και διάφορες ε, εταιρείε, ε, όπως είπε ο κ. Βασίτης, υποβάλλουν διαφορετικά στοιχεία. Ναι, υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη. Πολύ διαφορετική, πολύ διαφοροποιημένη συμμετοχή όταν πρόκειται για θέμα συνεργασίας με την Όλαφ. Ορισμένοι λένε ότι και μέσα στο ιστορικό κρατών μελών υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις μεταξύ των ε, υπηρεσιών ε, δικαιοσύνη, αστυνόμευσης, τελωνίων και των διοικητικών αρχών. Είναι λοιπόν δύσκολο, ίσως και όχι πολύ ενδιαφέρον, να πω αυτή η χώρα είναι πιο συνεργάσιμη από την άλλη χώρα δύσκολα τα πράγματα να πει κανείς κάτι τέτοιο. Το μήνυμα που προσπαθώ να μεταβιβάσω προ τα κράτη-μέλη είναι ότι εμείς ίσως είμαστε ένα θετικό στοιχείο για αυτούς, γιατί πολλές από τις μεγάλες απάτες γιατί πολλά τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο, όταν πρόκειται για μεγάλες απάτες δηλαδή. Και γι' αυτό όταν δεν παίρνουμε στοιχεία από τα κράτη-μέλη, λυπούμεθα. Και αυτό που θα ήθελα θα ήταν να έχουμε περισσότερα άτομα στην Όλαφ από εθνικές αρχές αστυνόμευσης. Μεταξύ 300 περίπου ερευνητών που έχω στην Όλαφ, δεν έχω κανέναν από τις γερμανικές υπηρεσίες αστυνόμευσης. Έχω από τα τελωνία. τελωνία ναι. Ούτε έναν όμως από την αστυνομία ή Bundeskriminalamt ή οτιδήποτε. Κανέναν από τις γαλλικές υπηρεσίες αστυνόμευσης. Ούτε έναν, ούτε έναν. Ε, δεν κατηγορώ εγώ τα κράτη-μέλη του εναντίον. Εγώ ως γενικός διευθυντής της όλα, θα πρέπει νομίζω να ανησυχώ γι' αυτό. Γιατί είδαμε και βλέπω με την πείρα που έχω μέχρι στιγμής, σας είναι και σύντομη, ότι εκεί, σε εκείνες τις χώρες που έχουμε, που έχουμε στην Όλαφ άτομα από τις Εθνικές Αρχές Αστυνόμευσης, βλέπουμε τι γίνεται. Έχουμε δηλαδή καλές πληροφορίες εκεί, καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Για προφανούς λόγους. Δεν διαμαρτύρομαι λοιπόν, θα ήθελα αλλά δεν το κάνω και για δύο λόγους. Ένα επειδή ανέφερε ο κύριος Γκάιερ γιατί δεν έχουμε πόρους και δεύτερον γιατί έχω μόνο τρεις από τις 500 θέσεις που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή στην Όλαφ. Τρεις λέω από 500. Δεν μπορώ λοιπόν να προσλάβω παρά μόνο τρία άτομα. Τι θα τα κάνω τα τρία άτομα. Uh, Τώρα, το άλλο θέμα για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι να αλλάξουμε τους δείκτες. Φοβούμαι ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε αργότερα, αλλά η έκθεση, όχι αυτή, αλλά η έκθεση για το άρθρο 325 για τις αντασταλίες και απάντες είναι σημαντικό θέμα αυτό. Και πολλές φορές μάλιστα παραπλανητικό θέμα, γιατί έχουμε ορισμένε χώρες που παρουσιάζουν πολλές ατασταλίες. Άλλες όχι. Και εργαζόμαστε σκληρά, ούτω ώστε όλα τα κρατημένη να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο, τα χρησιμοποιούν τα ίδια πρότυπα. Αλλά δεν είναι η δουλειά μας αυτή εμείς να τους κυνηγάμε. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τις εκθέσεις. Και όσο πιο καλές είναι αυτές οι εκθέσεις, τόσο πιο πολύ κατηγορούνται ότι είναι απαταιώνες. Και γι' αυτό υπάρχει η τάση των κρατών μελών να πούνε, κοιτάξτε, εμάς κατηγορείται επειδή υποβάλλουμε σωστές εκθέσεις. Ε, την επόμενη φορά δεν θα υποβάλλουμε. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η αριστερία δεν σημαίνει απάτη, απαραίτητο. Επίση, όπω είπε και ο κ. Βαλτσίτη, για τι έρευνε μα Έχουμε περισσότερε έρευνε σε ορισμένε χώρε. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητο ότι σε αυτές τις χώρες υπάρχουν περισσότερες απάτες. Ε, το θέμα είναι ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις χώρες. Μας δίνουν, δίνουν δηλαδή αυτοί περισσότερες πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, άμα κοιτάξετε τον πίνακα, βλέπετε και έχει μια στήλη που λέει καπνό ή τσιγάρα, δεν θυμάμαι τι λέει ακριβώς. Και υπάρχουν κάποιες έρευνες σε κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το κράτος μας έδωσε πληροφορίες οι υπηρεσίες τελωνίων μας έδωσε λέω πληροφορίες για λαθρεμπόριο καπνό. Και γι' αυτό κάνουμε την έρευνα εκεί. Δεν σημαίνει ότι εκεί υπάρχουν περισσότερες απάτες. Πράγμα ήταν αυτό βέβαια. Περισσότερες έρευνε σε μία χώρα μέλος σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες και περισσότερη συνεργασία. Αυτός δηλαδή ίσως είναι και ένας καλός δείκτης. θα ε, βελτιώσουμε τον τρόπο τον οποίο παρουσιάζουμε τα στοιχεία αυτά, θα αλλάξουμε λιγάκι τους πίνακες για να τονίσουμε περισσότερο το επίπεδο συνεργασίας των κρατών μελών. για να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη να συνεργάζονται μαζί μας και να έχουν καλύτερες διακρίσεις μεταξύ εκείνων των χωρών που υπάρχουν περισσότερες απάτες, πραγματικά, και εκείνες τις χώρες που συνεργάζονται περισσότερο από ό,τι άλλε μαζί μα για να καταπολεμήσουμε τις απάτες που υπάρχουν. Το τελευταίο θέμα του κυρίου Γκάιερ. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Πολλά προσπαθούμε να κάνουμε. Κυρίως να ορθολογικοποιήσουμε την χρήση των πόρων μας. Πρέπει να είμαστε βέβαια ρεαλιστέ. Και σκοπεύω να είμαι ρεαλιστή. Δεν θα συζητήσω περισσότερα χρήματα γιατί ξέρω ότι δεν θα μου δώσετε. Θα προσπαθώ να παραμείνω στο... στα χρήματα που έχω και ξέρω ότι ο υπερβολισμό μα ε, για πρώτη φορά περικόπη. Καλύτερη χρήση του προσωπικού. Όπως σας είπα θα πρέπει να κάνουμε διάκριση των διαφόρων αρμοδιοτήτων μέσα στο πλαίσιο της Όλαφ. Η Όλαφ έχει δύο έντολες. Η μία είναι γενική, έρευνες κατά της ε, απάτης. Ε, το άλλο είναι η πολιτική, γιατί είμαστε στην υπηρεσία της Κομισιόν για να προετοιμάζουμε την ε, πολιτική κατά των απατών. Και θα πρέπει βέβαια να χρησιμοποιούμε το προσωπικό ανάλογα. Μέχρι στιγμής καμιά φορά υπάρχουν επικαλύψεις, υπάρχουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και εξ αυτού και σπατάλη πόρων. Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου θα ξέρουμε, και αυτό νομίζω είναι ένα ερώτημα των υπηρεσιών που μας ελέγχουν, των σωμάτων που μας ελέγχουν και του κοινοβουλίου φυσικά, για το πόσα άτομα χρησιμοποιούνται για τις έρευνες αυτές. Και η απάντηση θα είναι πολύ πιο σαφής. Κάτι άλλο. Μειώνουμε το ύψος των πόρων που χρησιμοποιούμε για τη συνέχεια, όπως λέμε, που δίνεται. Που την 1η Φεβρουαρίου θα αποκαλείται η φάση της ε, εφαρμογής των συστάσεων της Όλαφ. Μετά που θα κάνουμε δηλαδή τις συστάσεις των Αρχές, ελέγχουμε και επιτηρούμε ή αν θέλετε βοηθάμε τις οικονομικές ή δικαστικές αρχές στην εργασία τους. Καμιά φορά έχουμε καμιά εκατοστή δικαστικές περιπτώσεις. Εκατοντάδες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, από την Ούκλαφ. Με δικαστική συνοχή. Υποθέσεις που δεν τις γνωρίζει κανένας. Και υπάρχουν σε κάποια αρχεία, σε κάποια χρονοτούλαπα εκεί στην Κομισιόν. Και θα χρησιμοποιούμε καλύτερα τους κόσμους, θα έχουμε λιγότερα άτομα που θα ασχολούνται με το θέμα αυτό, αλλά θα ασχολούνται πιο αποτελεσματικά και περισσότερους που θα κάνουν τις πραγματικές έρευνες. Δηλαδή θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουμε, κυρίως δηλαδή τις έρευνες και σε άλλες μονάδες ασχολούνται με την πολιτική κατά της απάτης και λιγότεροι που θα ασχολούνται με τις επαναλαμβανωμένες επαναλαμβανομένες ε, διοικητικές εργασίες. Τέλος, όσον αφορά τους περιορισμένους πόρους, το ετήσιο πρόγραμμα που τελειοποιείται αυτές τις μέρες θα δίνει πιο ξεκάθαρα μηνύματα όσον αφορά τις προτεραιότητες, ιδίως για τις έρευνες. Εγώ προτρέχω λίγο αυτό που θα υπάρχουν στον κοινό κανονισμό που συζητάτε που θα πρέπει να καθορίζει τις προτεραιότητες στην επιλογή των υποθέσεων στη φάση δηλαδή την εμπλεκτική των ερευνών και θα αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της διαφθοράς και του οργανωμένου κλίματος που είναι πολύ πιο δύσκολο να τα βρούμε. Και επίσης θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποιους γεωγραφικά επικίνδυνους τομείς όπου θα ανοίξουμε περισσότερε έρευνε. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρέσλε, ευχαριστώ. Μία ερώτηση μόνο ήθελα να κάνω. Τι πιστεύετε κύριε Γενική Διευθυντά για τη φήμη ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η δυνατότητα πρόσληψη προσωπικού σε ό,τι αφορά το AIPN. Αυτό ισχύει ή όχι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Ανησυχώ κάπως, γιατί άκουσα και δεν θυμάμαι καν πού και από ποιον και σε ποια περίσταση, σε ποια καντίνα το άκουσα, σε ποια κηλικία το άκουσα. Εδώ στο κοινοβούλιο. Ανησυχώ γιατί δεν έχω σχετικές πληροφορίες. Αλλά φαντάζομαι ότι αν δεν αλλάξετε τίποτα, δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Πιο πολύ από το δικό σας χέρι περνάει παρά από το δικό μου. Άρα η απάντησή μου δεν αλλάζει κάτι. Αν συμφωνείτε και εσείς ασφαλώς. Συμφωνείτε, πολύ ωραία. Μάλιστα. Τότε αισθάνομαι και εγώ ασφαλής. Κανείς άλλος. Ο κύριος Παλσίτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, όπως είπατε, ορθώς πολλά θα πρέπει να αλλάξουν. Και νομίζω ότι η έκθεση αυτή, αυτόν τον σκοπό ακριβώς θα εξυπηρετήσει στο μέλλον, σε ό,τι αφορά τις αρχές μας και τους τομείς δραστηριότητά μας. Μελλοντικός μας στόχος είναι να μην δημιουργούνται τόσο πολλές ε, έρευνες, αλλά αφετέρου μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μαζί με την ανεξάρτητη όλα θα πρέπει να θέσουμε και να καταρτήσουμε μια πολιτική κατά της απάτης και να υπάρχει και εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής αυτής. Θα πρέπει να υπάρχουν και να διενεργούνται, βασικός μας στόχος αυτός είναι, όσο το δυνατόν λιγότερες έρευνες γίνεται και μόλις εφαρμοστούν οι πολιτικές αυτές, θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι. Σήμερα ακούσαμε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία είναι πιο διατεθειμένα να συνεργαστούν με την Όλαφ παρουσιάζουν χειριχεία. Άρα θεωρώ ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί βασική κατευθυντήρια γραμμή στο μέλλον. Και εσείς θα πρέπει να μας πείτε πώς θα εφαρμοστεί το σύστημα προκειμένου να έχετε επαρκή στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη. Προκειμένου η τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των ε, κοινοτικών πόρων, να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να δώσουμε σαφείς απαντήσεις στους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις ε, εκτενείς απαντήσεις σας και προστοκούμε και στις ε, περαιτέρω συζητήσεις και ελπίζουμε η τρέχουσα μεταρρύθμιση που συζητήσαμε και το πρωί να διευκολύνει το έργο σας και το δικό μας, τη δική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Merci. Interventions? Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις. Όχι. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο, οπότε προτείνω να κλείσουμε την Εξέταση του σημείου 7 για την ετήσια έκθεση 2011 που αναφέρεται στο 2010. Να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Διευθυντή Κέσλερ καθώς και τους συνεργάτες του και να περάσουμε στην εξέταση του σημείου 8 που είναι η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου με τίτλο «Έλεγχος της διαδικασίας ακαθάρισης λογαριασμών». Χαιρετίζω τους τον κύριο Μισελ Κρετά που είναι εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου απόψε και την εισηγήτρια κυρία Γκρέσλε και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου για να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματά του. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η έκθεση που σας υποβάλλω σήμερα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εξετάζει τη λειτουργία της διαδικασίας εκαθάρισης λογαριασμών στον τομέα της γεωργίας και των φυσικών πόρων για τους οποίους η Ένωση δαπανά ετησίως γύρω στα 55 δις ευρώ. Τι είναι η εκαθάριση λογαριασμών. Πρόκειται για μια διαδικασία που ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης και που αφορά συγκεκριμένα τις δαπάνες που έχουν εκτελεστεί στην διαχείριση Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να μπορέσει η Επιτροπή που δεν εκτελεί άμεσα αυτές τις δαπάνες να αναλάβει την τελική της ευθύνη στην εκτέλεση του προπολογισμού και συγκεκριμένα εξασφαλίζοντας ότι η δαπάνη ήταν σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό μας εξηγεί το άρθρο 53 ε, του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Αυτή η διαδικασία εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στο πρώτο στάδιο η ε, Κομισιόν λαμβάνει την απόφαση δημοσιονομικής εκαθάρισης μέσω της οποίας εκφράζεται για την ακρίβεια των λογαριασμών που τις έχουν ε, κοινοποιήσει οι υπηρεσίες ε, πληρωμής των κρατών μελών. Για να λάβει αυτή την απόφαση στηρίζεται στους εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης που πιστοποιούν τους λογαριασμούς αυτών των ε, υπηρεσιών καταβολής των πληρωμών. Σε δεύτερη φάση, η ίδια η Κομισιόν προβαίνει σε ελέγχους ώστε να εντοπίσουν και να αποκλείσουν ε, χρηματοδότη τις ε, δαπάνες που δεν είναι σύμμορφες με τους κοινοτικούς κανόνες. Αυτή η δεύτερη απόφαση ονομάζεται η απόφαση ε, συμμόρφωσης. Στην παρουσία μου αυτή θα μιλήσω πρώτα για την εκαθάριση λογαριασμών, έπειτα την εκαθάριση λογαριασμών ως προς τη συμμόρφωση και έπειτα για τη διαδικασία εκαθάριση λογαριασμών συνολικά, δηλαδή εξετάζει συνολικά τα δύο είδη απόφασης για τις οποίες σας ε, μίλησα ήδη. Καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι παρατηρήσεις του συνεδρίου δεν είναι νέες και έχουν ήδη υποβληθεί είτε σε αιτήσεις εκθέσεις είτε μέσα σε ειδικέ εκθέσεις. Αντίθετα, η συγκέντρωση αυτών των παρατηρήσεων σε ένα συνεπές και ομοιόμορφο πλαίσιο επιτρέπει να έχει κανείς μια γενική εικόνα. Και αυτό είναι κάτι νέο σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, η δημοσιονομική εκαθάριση λογαριασμών. Εν γέννη, και παρά δυναμίες για ορισμένα σημεία που αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση και από τον οποίο δεν θα επεκταθώ εδώ, το συνέδριο διαπίστωσε ότι η εργασία των οργανισμών πιστοποίησης επιτρέπει στην Κομισιόν να έχει επαρκείς πληροφορίες και ε, αξιόπιστες στη διάθεσή της για να προβεί στην ετήσια απόφασή της για δημοσιονομική καθάριση λογαριασμών. Ωστόσο, από το 2007 οι εργασίες αυτών των οργανισμών πιστοποίησης έχουν επεκταθεί σε ορισμένες πτυχές της νομιμότητας και της κανονικότητας των πληρωμών για με τις οποίες δεν ασχολούνται στο παρελθόν. Και το συνέδριο διαπίστωσε πως αυτά τα νέα καθήκοντα δεν ήταν απόλυτα υποέλεγχο από πλευράς των οργανισμών πιστοποίησης. Εν γέννη, η προστιθέμενη αξία της νομοδότησης που εκφέρουν αυτοί οι οργανισμοί για τη δήλωση αξιοπιστίας των διευθυντών των υπηρεσιών καθάρισης δεν είναι ακόμα εμφανής αυτή η προστιθέμενη αξία. Κατά δεύτερο λόγο, ε, μάλλον δεύτερο είναι η εκαθάριση λογαριασμών ως προς τη συμμόρφωση που παρέχει στην Κομισιόν μια σημαντική αρμοδιότητα. Από το 1999 μέχρι το 2010 η Κομισιόν έχει αποκλείσει από τους λογαριασμούς του, της Ένωσης ένα ποσό άνω των 6 δις ε, πέρα από τις, ε, που αφορούν μάλλον παρατυπίες δαπανών. Ωστόσο, το συνέδριο διαπίστωσε ότι αυτή η εκαθάριση λογαριασμών ως προς τη συμμόρφωση γινόταν με κάποιο τρόπο που παρουσιάζει κάποια προβλήματα, εκ των οποίων θα αναφέρω τρία. Πρώτον, η περιορισμένη πόροι που έχει στη διάθεσή της η Κομισιόν για να προβεί σε αυτούς τους ελέγχους συμμόρφωσης και η μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιεί για να επιλέξει τους τομείς ε, επί των οποίων εστιάζει την προσοχή της δεν της επιτρέπουν να καλύψει με ικανοποιητικό τρόπο το σύνολο των γεωργικών δαπανών. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι υποτομείς που διαφεύγουν. Δεύτερη παρατήρηση για τη συμμόρφωση τα ποσά των δαπανών που αποκλείονται από την κοινοτική χρηματοδότηση μέσω των αποφάσεων συμμόρφωσης προκύπτουν κατά βάση, δηλαδή πάνω από το 90% αυτών, προκύπτουν από ε, καταποκοπήν ε, διορθώσεις. Ε, αυτά τα ποσά υπολογίζονται από τις υπηρεσίες της Κομισιόν επί τη βάση των ανεπαρκειών που έχουν διαπιστώσει στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Δεν βασίζονται στα ποσά των σφαλμάτων στις πληρωμές που έχουν καταβληθεί στους τελικούς δικαιούχους της ε, βοήθειας, της ενίσχυσης. Προκύπτει λοιπόν ότι αυτές οι ε, κατά αποκοπήν διορθώσεις δεν αντιστοιχούν σε ένα μέσο διόρθωσης των παράνομων πληρωμών. Αντίθετα, είναι πολύ χρήσιμες για να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το συνέδριο εδώ και καιρό έχει ε, σημειώσει αυτή τη δυσκολία και θα θυμίσω πως αυτή η παρατήρηση ήδη είχε ληφθεί υπόψη από το Ευρωκοινοβούλιο στο ψήφισμα απαλλαγής για τους λογαριασμούς του 2007 όπου το Ευρωκοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το ότι καμία ε, έγκυρη συσχέτιση δεν μπορούσε να υπάρχει ανάμεσα στις λογιστικές διορθώσεις και τα πραγματικά ποσά αντικανονικών πληρωμών. Τρίτη αδυναμία, την οποία έχει εντοπίσει το συνέδριο, οι αποφάσεις συμμόρφωσης υιοθετούνται πολύ αργά. Επιπλέον, η παρέμβαση μιας διαδικασίας συνδιαλλαγής ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κρατη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρατείνει την προθεσμία υιοθέτηση αυτών των αποφάσεων συμμόρφωσης. Αυτές οι χρονικές ε, προθεσμίες ε, είναι της τάξης των τριών ε, με πέντε ετών και κάποιες φορές και παραπάνω. Και για παράδειγμα ε, το συνέδριο υπογραμμίζει το γεγονός ότι στο τέλος του 2008, επί των οποίων τον οποίο αφορούν οι παρατηρήσεις μας, η καθάριση των λογαριασμών δεν είχε ολοκληρωθεί για καμία χρήση μετά το 2001. Δηλαδή, στο τέλος του 2008, η τελευταία χρήση για την οποία είχε γίνει η εκαθάριση των λογαριασμών ήταν το 2001. Τρίτο σημείο και διατυπώνω εδώ κάποια συμπεράσματα για τη διαδικασία καθάρισης εν γέννη. Δηλαδή, ε, εξετάζοντας τα δύο είδη ε, ε, απόφασης, τα οποία σας ανέφερα χωριστά. Θα έχω να κάνω εδώ λοιπόν τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, το συνέδριο διαπιστώνει ότι στο τέλος της σημερινής διαδικασίας η Κομισιόν δεν λαμβάνει απόφαση ορίζοντας με τελεσίδικο τρόπο και για συγκεκριμένη χρήση τα ποσά των γεωργικών δαπανών που αναγνωρίζει ότι βαραίνουν επιβαρύνουν τον προπολογισμό της Ένωσης. Όμως, κανονικά, αυτό λέει ο δημοσιονομικός κανονισμός, στο άρθρο 42 του διαδικαστικού κομματιού αυτού του κανονισμού ορίζει ότι η διαδικασία καθάρισης προβλέπει τον καθορισμό από πλευράς Κομισιόν του ποσού δαπανών που θεωρείται ότι επιβαρύνει τον προπολογισμό. Τη απουσία αυτής της οριστικής απόφασης η πληροφορία αυτή, δηλαδή το ποσό των δαπανών που ορίζεται τελεσίδικα ότι επιβαρύνει τον προπολογισμό, αυτή η πληροφορία δεν συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα απαλλαγή διατυπώνει μια γνωμοδότηση για τις... Ε, για τις διαδικασίες επί των οποίων η Κομισιόν δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη για τα ποσά που παρουσιάζονται στους λογαριασμούς μπορεί να αλλάξουν, να τροποποιηθούν μετά την απαλλαγή όταν θα γίνουν οι καθαρίσεις συμμόρφωση τη επιτροπή. Δηλαδή η απαλλαγή αφορά ένα ατελές έγγραφο. Τρίτον, διαπιστώνει επίσης το συνέδριο ότι για τις ε, καταποκοπήν διορθώσεις. Η επιβάρυνση οικονομική στην ουσία βαραίνει τα κράτη-μέλη. Τα κρατη και όχι τους δικαιούχους της βοήθειας που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. Με, παρά αυτόν τον ε, χαρακτήρα των καταποκοπήν δεν συνδέεται αυτό άμεσα με τι ε, αντικανονικότητε, τι παρατυπίε που έχουν διαπιστωθεί και μάλιστα πολλέ από αυτέ τι υποθέσει βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και από την άλλη πλευρά, επειδή τα ποσά αυτά πληρώνονται από του φορολογούμενου και όχι από του δικαιούχου των ε, ενισχύσεων, αυτέ οι επιστροφέ τι οποίε απαιτεί, οι αποζημιώσει, μάλλον που απαιτεί η Κομισιόν δεν έχουν το αποτέλεσμα το αποτρεπτικό ούτε το διορθωτικό για του λογαριασμού. Ολοκληρώνω θυμίζοντας τις συστάσεις του συνεδρίου για αυτά τα σημεία και θα τα αναφέρω πολύ σύντομα, συνοψίζοντας. Ε, το συνέδριο διατυπώνει δύο βασικές ε, συστάσεις. Ε, καταρχήν, συστήνει να διευκρινιστούν οι στόχοι των διαφορών φάσεων της διαδικασίας καθώς και ο ρόλος των διαφόρων μπλεκόμενων μερών σε αυτές τις διαδικασίες και πιο συγκεκριμένα συστήνει τη θέσπιση προθεσμιών για την εκτέλεση των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας έτσι ώστε να γίνει μια προσπάθεια μείωσης της ε, διάρκειας αυτής της διαδικασίας. Έπειτα συστήνει η Κομισιόν να ορίσει με μια τελεσίδικη απόφαση τα ποσά δαπανών που ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη οικονομική χρήση. Το, η Κομισιόν να συμπεριλαμβάνει τα ποσά αυτά στους λογαριασμούς της συγκεκριμένης χρήσης και να ενημερώνει και την αρχή αρμόδια για την απαλλαγή, ώστε αυτή να μπορεί να αποφασίσει εν πλήρη γνώση των, των όλων των λεπτομεριών. Αυτά ε, έχω να πω. Ε, για να συντομεύσω την εισήγησή μου, αλλά δεν θα ήθελα να κλείσω χωρίς να ευχαριστήσω την εισηγήτριά σας και τους συνεργάτες σας για το ενδιαφέρον που έδειξαν για το θέμα αυτής της έκθεσης, καθώς και για την ποιότητα της συνεργασίας που χαρακτήρισε την συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια Ίγκα έχει λόγο. Μάλιστα τόσο πολύ έκτακτη έκθεση που δεν μπορούσα να την αφήσω από τα χέρια μου. Είναι μια έκθεση που παρουσιάστηκε πέρσι και το γεγονό ότι την εξετάζουμε μόλι σήμερα είναι ότι μετά από την προσεκτική ανάγνωση τόσο σημαντική και ενδιαφέρουσα αυτή τη έκθεση, αποφάσισα να περιμένω την εξεργασία μέχρι να έχουμε και μια νέα έκθεση, έκτακτη έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου, όσον αφορά την ε, επανάκτηση αχρηστήτως καταβεβλημένων ποσών. Το Σκύτο το είπε, έχουμε ένα πολυσχηδές ε, πρόβλημα που αφορά άμεσα τον έλεγχο του προπολογισμού. Είναι μια έκθεση ουσιαστική και βασική σημασία για την εργασία μα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται σε μια διεθνή επιχείρηση όταν δώσει την απαλλαγή στο Προεδρείο η Γενική Συνέλευση και μετά πρέπει να διορθωθούν τα αριθμητικά στοιχεία. Αυτό μα συμβαίνει εμά κάθε χρόνο χωρί να μα απασχολεί. Περί αυτό πρόκειται και προσπάθησα γι' αυτό να υποβάλω προτάσει πώ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η διόρθωση των αριθμητικών στοιχείων. Ο καθένας μας ξέρει ότι το πρόβλημα που σημειώνει το ελεκτικό συνέδριο, δηλαδή εκ των υστέρων αυτές διορθώσεις και το ότι τα στοιχεία, η, τα βιβλία είχαν κλείσει μέχρι το 2001, ότι αυτό βασίζεται κατά βάση στους ίδιους τους κανονισμούς. γιατί ελέγχουμε στον αγροτικό τομέα τον έλεγχο μόνο του 5% των δαπανών. Και για το 5% αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Διόρθωση του 100% βέβαια δεν είναι κάτι που θα μπορεί κανένας να λάβει υπόψη. Και θα πρέπει κατά βάση να έχουμε περισσότερα στοιχεία στα χέρια μας. Γι' αυτό ακολούθησα όλες τις ε, προτάσεις του Ελεκτρικού Συνεδρίου γιατί ελπίζουμε να έχουμε έτσι καλύτερη βάση στοιχείων. Και κάθε εισηγητή για την απαλλαγή θα πρέπει να έχει ένα κεφάλαιο που να αφορά αυτές τις εκ των διορθώσεις των ετησίων λογαριασμών. Προσπαθώντας να τις αντικατοπτήσει σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Αυτό θα ήθελα να κάνει το σώμα τουλάχιστον. Αυτό το έργο του 5% και η προβολή στο 100% δεν είναι πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι βέβαια και το γράφει το συνέδριο ε, ξεκάθαρα είναι ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα στοιχεία που δίνουν το κράτη Δηλαδή εκεί υπάρχει κάποια αβεβαιότητα, κάποια ασάφεια και δεν μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση και υπάρχουν γι' αυτό διάφορες τροπολογίες ότι προσπαθούμε ακριβώς να λύσουμε αυτό το θέμα. Πώς μπορούν δηλαδή οι αρχές ελέγχου επιτόπου να είναι πιο αποτελεσματικέ τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να βασίσουμε καλύτερα στα στοιχεία τους. Γιατί τι να κάνω μια εθνική δήλωση που να βασίζεται να ελευθερώνει σε ασφαλμένα στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εκπαιδεύσουμε τα κράτη-μέλη. Και τώρα αναφέρω αυτό στο σημείο 3 της τυχής μου έκθεση και υποβάλλω και κάποιες προτάσεις πώς μπορούμε να διορθώσουμε. Και μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Εκτελεστική Επιτροπή εδώ να αναφερθεί στα κράτη-μέλη για άλλη μια φορά και σε όλα τα προβλήματα που βλέπουμε επί τόπου και που γνωρίζουμε βέβαια βαρκώς αν δεν τα καταφέρουμε στον αγροτικό τομέα όπου είναι αρκετά σαφή η κατάσταση δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε με θέση μία. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο αγροτικός τομέα. Όσον αφορά τα κεντρικά προβλήματα των έλεγχων του 5% και της ποιότητας των αρχών επιτόπου, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα τα ανεπαρκή συστήματα της ε, ανάξιων των Και αυτά που είπε ο κύριος Κρετέ μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλά παρουσιασμένα γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια ανέκτησε η Κομισιόν 5-6 δισεκατομμύρια. Για να δούμε τώρα. Στα 17 χρόνια δαπανήθηκαν 500 δισεκατομμύρια, ανακτήθηκαν όμως κάπου ε, το 1%. Δηλαδή το σύστημα μας ε, προβλέπει ότι είναι πιο ακριβό να γίνονται οι έλεγχοι παρά να καταβάλλονται κάποια χρεωστήτα ποσά. Άσχετα τι θα κάνουμε δηλαδή. Σε καλύτερη περίπτωση Έχουμε πολύ λυπηρή κατάσταση στην αγροτική πολιτική και δύσκολη. Δεν θέλω να προκαλέσω την Κομισιόν. Θέλω να πω ότι κάναμε μια σειρά συνεδριάσεων και δεν καταφέραμε όμως να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Δεν θέλουμε βέβαια να επιβάλλουν περισσότερη γραφειοκρατία, αλλά θα ήθελα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα επί τόπου, τάπτω, συγγνώμη, θα να τα εξετάσουμε καλύτερα. Και αυτό η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ καλή μου φαίνεται, για την εκαθάριση των λογαριασμό. Θα πρέπει να εξετάσουμε όμω πώ θα έχουμε πιο ακριβεί και πιο καλέ πληροφορίε και προ όφελο προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση. Αυτά είχα να πω και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση με τους βουλευτές. Αλλά προηγουμένως μήπως η Κομισιόν θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Καταρχάς, κυρίες και κύριοι βουλευτές και κύριοι Κροτάν, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε για να μιλήσω σήμερα για τα θέματα αυτά, γιατί θεωρώ ότι η δική έκθεση και το έγγραφο εργασία της κυρίας Γκρέσλε αποτελούν μια πολύ καλή βάση. Συμφωνούμε με την απόψη της κυρίας Γκρέσλε ότι δεν είναι, ε, δεν συστήνεται με τους ε, σημερινούς όρους μεταρρύθμιση βασική του συστήματος. Αυτό αξιολογήθηκε. Η κοινή γεωργική πολιτική επί σειρά ετών έχει περίπου 2% ποσοστό σφαλμάτων. Και αυτό κυρίως για τον πρωτοπυλώνα που αποτελεί το μερδί του λέοντος και είναι λίγο λιγότερο από 2%. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα για τα αριθμητικά στοιχεία ως προς τον έλεγχο που αναφέρθηκαν η κυρία Γκρέσλε. Ίσως θα μπορέσουμε να βρούμε έτσι μια κοινή βάση. 5% των ταπανών, είπατε, ε, ελέγχονται. Και αυτό το προβάλλουμε στο 100%. Αλλά στα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι όλες οι αιτήσει ελέγχονται ε, από διοικητικής άποψης και έχουμε ελέγχου επιτόπου σε ύψο 5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει με τη σειρά της το έργο των κρατών μελών και περίπου 50% των δαπανών ανά έτος ελέγχονται. Άρα θα δημιουργούταν λάθος εικόνα αν λέγαμε ότι μόνο 5% ελέγχεται και ότι αυτός είναι όλος ο έλεγχος για τα 55-85 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Πιστεύουμε ότι γι' αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και να εξελιχθεί το σημερινό σύστημα και καταθέσαμε σχετικές προτάσεις για μια νέα, ένα νέο οριζόντιο κανονισμό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 10 Οκτωβρίου στα πλαίσια της μεταρρύθμισης ΚΑΠ. Δύο από τις βασικές συστάσεις περιλαμβάνονται στο σημείο 1 του εγγράφου εργασίας. Όντως είναι επιθυμητό η διάρκεια των διαδικασιών συμμόρφωσης να μειωθεί κατά το δυνατό. Και έτσι σε αυτό προσανατολίζονται και τα σχέδια για τους ε, ελέγχους μας και η χρήση των πόρων μας. Οι πόροι αυτοί ασφαλώς και είναι περιορισμένοι για το ποσό των 55 δισεκατομμύριο έχουμε περίπου 220 άτομα που εμπλέκονται με οποιαδήποτε μορφή με τον έλεγχο. 10% περίπου του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Ωστόσο, αμφιβάλλουμε κατά πόσον ε, η εισαγωγή νομικά δεσμευτικών ε, χρονοδιαγραμμάτων θα ήταν θεμητή. Θεωρούμε ότι αυτό θα ήταν ε, αντιφατικό με την πολυπλοκότητα κάποιων υποθέσεων και με το προϋπολογισμό κάποιων κρατών μελών και, τον και με τους περιορισμένους πόρους. Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί τα κράτη-μέλη, τα οποία συχνά είναι μικρά κράτη-μέλη και κράτη-μέλη με περιορισμένη διοικητική ικανότητα, θα πρέπει να προσέξουμε να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα υπεράσπιση του. Από αυτό εξαρτάται βασικά η ποιότητα τη διαδικασία και η αποδοχή του αποτελέσματος, τελική ανάλυση. Υποστηρίζουμε ωστόσο τη σύσταση τη κυρία. Ε, Γκρέσλε για τη διαδικασία ετησίας. Αυτή η διαδικασία σε 28% των περιπτώσεων οδήγησε σε διόρθωση 10%, 13% ήταν κάτω από 10% και σε άλλες περιπτώσεις, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι διορθώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, ήταν πιο περιορισμένε. Είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Άρα ελέγχουμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό με καλύτερη και με μεγαλύτερη ε, αποδοτικότητα. Το θέμα είναι να βρούμε το σωστό χρονικό σημείο στη διαδικασία συμμόρφωσης που μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία διατησία. Ε, αυτό σημαίνει, η διατησία σημαίνει ότι έχουν παγιωθεί οι δύο αντιφατικές θέσεις. Για τη δεύτερη σύσταση, στο σημείο 1 του εγγράφου εργασία. Μιλάμε για τη σύνδεση μεταξύ του ποσού του, της διόρθωσης και της έκτασης των ε, μη κανονικών πληρωμών. Και αυτό σημειώνεται ε, με κριτική διάθεση, αλλά θεωρούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όπως παρουσιάζονται στην ειδική έκθεση σε ό,τι αφορά τις εδαφικές επιδοτήσεις είναι δυνατόν όντως ε, να υπάρχουν απώλειες, ε, να υπολογιστούν οι απώλειες σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και μάλιστα με βάση τα ενημερωμένα στοιχεία και συστήματα εντοπισμού των ε, επιφανειών εκμετάλλευσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να υπολογίσουν το ύψος των διορθώσεων. Αυτό ε, προϋποθέτει ότι τα σώματα πιστοποίησης ε, μπορούν να ελέγξουν τα στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών και γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία και όταν η προστοποιούσα αρχή επιβεβαιώσει τα στατιστικά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί στην περίπτωση αυτή να ορίσει το αντίστοιχο ποσοστό σφάλματος και το σύστημα επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι ένα διοικητικό σφάλμα, για παράδειγμα, ε, είχε ως αποτέλεσμα τόσες ε, ε, λανθασμένες, τόσες μη κανονικές πληρωμές σε ό,τι αφορά τις επιστροφές. Είπατε ότι το ποσοστό των επιστροφών ήταν περίπου 1,5%. Θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν είναι κάθε αντικειπτικό σφάλμα συνδεδεμένο με λανθασμένες πληρωμές. Σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρχουν και λανθασμένες πληρωμές που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε επιστροφές γιατί δεν ήταν υπεύθυνοι οι γεωργοί και προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο, και εδώ επανέρχομαι σε κάτι που αναφέρεται στο έγγραφό σας κυρία Γκρέσλε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξαρτήσει τις διορθώσεις από τις διαπραγματεύσεις από τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης για τις διορθώσεις αυτές, ε, το ύψος ε, αυτό θα πρέπει να οριστεί η βάση του ποσοστού σφάλοντος. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε. Για το σημείο 2 της σύστασης τώρα που μιλάει για απαιτήσει για μεγαλύτερη διαφάνεια στην διαδικασία απαλλαγής. Να υποδείξω το εξής, ότι στη δεύτερη παύλα ήδη διατύφονται ε, οι απαραίτητες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση για συγκεκριμένα λογιστικά έτη. Θα ήθελα να σας πω να σας παραπέμψω στο σημείο 35 της έκθεσης ε, του 2010, όπου αναφέρεται ποια απόφαση ε, αναφέρεται και για ποιο λογιστικό έτος. Αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι η κατάσταση για την πρώτη και την τρίτη παύλα. Ζητούνται εκεί σε ό,τι αφορά τις διορθώσεις που βρίσκονται υπό, διαπραγμα... υπό εξέταση, υπό επεξεργασία. Θα πρέπει να πω ότι ήδη υπάρχουν στοιχεία για αυτά και στο σημείο 6 της αιτήσης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2010 για παράδειγμα. Τα στοιχεία αυτά, και αναφέρω το έγγραφο, να δίδονται στοιχεία κράτος μέλος και ανα έτος, θεωρούμε ότι δεν είναι εφικτή. Και γιατί, γιατί η διόρθεση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας συμμόρφωσης πρόκειται για ένα κινούμενο στόχο θα ήταν επιβλαβές για την λειτουργία της διαδικασίας και της λειτουργίας με το κράτος μέλος να δημοσιεύονται τέτοια στοιχεία πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες και τις ανώτατες τιμές θα έδινε ένα χαρακτήρα διαπραγμάτευσης ε, στη διαδικασία την οποία δεν δέχεται ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις, θέλουμε αντικειμενικά κριτήρια και η διαδικασία συμμόρφωση. Ε, άλλωστε δεν ε, λειτουργεί με ανώτατε και κατώτατε ε, τιμέ. δεν είναι αυτή η τεχνική που χρησιμοποιούμε, όχι. Ε, θα πρέπει να αξιολογηθούν αντικειμενικά τα σφάλματα. Τέλος, πώς θα πρέπει να μιλήσουμε για ελέγχους που ενδεχομένως να διεξαχθούν στο μέλλον, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πρέπει να διεξαχθούν ή θα μπορούν να διεξαχθούν. Επί ποιας βάσης θα πρέπει να βασιστούμε εδώ θα κάνουμε κάποιες εικασίες ε, και νομίζω ότι αυτό δεν εμπίπτει στο πλαίσιο μιας διαφανούς πολιτικής, στο πλαίσιο της απαλλαγής. Το τι δεν την παύλα να περάσω τώρα, επιτρέψτε μου. Μου φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό ο αριθμός να οριστεί ο αριθμός των περιπτώσεων που δεν ε, ακολούθησαν τη διαδικασία συμμόρφωσης. περίπου 50% σε μακροχρόνιο πλαίσιο και μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια προβολή. Ο λόγος είναι μάλλον απλός ότι οι ελεγχόμενες υποθέσεις ε, ελέγχονται σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για τον προϋπολογισμό. Δηλαδή το κομμάτι που δεν ελέγχεται έχει πιο χαμηλό ε, επίπεδο κινδύνου και άρα ε, επίπεδο σφάλματος. Δεν έχουμε τέτοια βάση λοιπόν για να γίνει τέτοια προβολή. Τώρα πόσες διορθώσεις γίνονται δεν μπορούν να γίνουν για, λόγω του, της περίοδου των 24 μηνών. Ούτε αυτό μπορούμε να το ορίσουμε. Μιλάμε για την επιστολή προς τα κρατημέλια που περιγράφεται ενδεχόμενο του σφάλμα τέτοιες δαπάνες δεν μπορούν να ελεγχθούν καθότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο νομικά. Ο κανονισμός προβλέπει οι δαπάνες οι οποίες είναι πιο παλιές από ότι 24 μήνες να παραμένουν κλειστές για ενδεχόμενους ελέγχους. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια στοιχεία. Αν το προσπαθούσαμε αυτό, θα κάναμε ε, επαχθείς εικασίες σε ό,τι αφορά σε τους σπόρους αυτούς που διαθέτουμε και οι πόροι αυτοί δεν υπάρχουν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διαβεβαίσω την κυρία Γκρέσλε ότι ιδιαίτερα επικίνδυνοι τομείς εξετάζονται εντελεχώς και προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται συχνά επισκέψεις έλεγχου, επιθεωρήσεις για να καλυφθούμε σε αυτούς τους τομείς υψηλής επικινδυνότητας σε ό,τι αφορά τις ε, συστάσεις στο σημείο 3 για την διαχείριση των ελέγχων. Υπάρχει ήδη ένα σύστημα το οποίο δίνει πρόσβαση στο σύστημα RIPAC στα κρατη το οποίο έχει περάσει και σε υπολογιστικά συστήματα πλέον, σε ό,τι αφορά τα πρίμια της επιχειρήσης στα κράτη-μέλη. Επίσης ελέγχουμε δυνατότητες για την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των επιστοποιούσεων αρχών. Αυτό γίνεται με βάση μια αξιολόγηση κινδύνου ύστερα σε ό,τι αφορά την βελτίωση της ε, δηλώσης αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τις αρχές αυτές πιστοποίησης. Το εξετάσαμε και αυτό το θέμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόταση, ο πρόταση για ε, οριζόντιο κανονισμό προβλέπει τέτοιους, ε, τη μείωση τέτοιων επιτόπιων ελέγχων στα κράτη-μέλη, αν διαθέτουν συστήματα καλού ελέγχου και έτσι το ποσοστό σφάλματος έχει ένα αποδεκτό επίπεδο συνεργαζόμαστε με τις ε, επιτόπιες αρχές, με τις υπηρεσίες αυτές, για να μπορέσει να καταστεί λειτουργικός ο κανονισμός αυτός. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά αυτός ο στόχος, αυτός είναι ο απότερος στόχος, γιατί αυτό καθιστά σαφές ότι στην τελική ανάλυση το θέμα είναι να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι φυστάμενοι πόροι για τον έλεγχο. Και γι' αυτό λοιπόν τα κρατημέλη τα οποία εργάζονται πάρα πολύ καλά και που παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο σφάλματος θα πρέπει να έχουν ένα πλεονέκτημα για τη διεξαγωγή λιγότερων επιτόπιων ελέγχων. Τώρα η ανάλυση της ορθότητας των δηλώσεων αξιοπιστίας. Αυτό γίνεται στη Γενική Έκθεση Δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά το επίπεδο σφάλματος, να σας παραπέμψω στην παράδειγμα 7 της έκθεσης αυτής. Για κάποιες τις συστάσεις στο σημείο 3 παρουσιάζονται κάποια προβλήματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Αυτό ισχύει καταρχάς ε, για την εκπαίδευση εθνικών αρχών, εθνικών υπαλλήλων, ε, κατάρτιση αυτό κανονικά δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο σε διάφορες συναντήσει προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή προκειμένου να διαβιβάσουμε τα στοιχεία εκείνα, τη γνώση εκείνη που χρειάζεται για να γίνεται σωστά το έργο, να επιτελείται σωστά το έργο σε ό,τι αφορά τους ε, εθνικούς υπαλλήλους ε, και το δεν θα πρέπει να τιμωρούνται όταν ανακαλύπτουν λάθη, ασφαλώ αυτό δεν ε, αποτελεί κάτι το οποίο είναι στην ευκαιρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι άλλο τώρα, να ευχαριστήσω και την κυρία Γκρέσλα και το Ελεκτικό Συνέδριο για την Ηθική Έκθεση. Θα λάβουμε πολύ στα σοβαρά τι συστάσει αυτέ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμοστούν εφόσον περνάει από το χέρι μα και ασφαλώ ε, θα συζητήσουμε τι διάφορε συστάσει. και όπου ενδεχομένως υπάρχουν παρανοήσεις ε, ασάφειες θα προσπαθήσουμε μέσω συζήτησης να και διευκρινίσουμε. Merci, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μέπλε. Εντάξει, το πρόεδρο μα του Σκοκομπιού έφτασε και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και μετά θα ξαναδώσω την Προεδρία. Μπορεί να αρχίσει η συζήτηση τώρα. Η κυρία euh, ε, θέλει ίσως ε, το ηλεκτρικό συνέδριο να δράσει σε αυτά που είπε η Επιτροπή. Για να τα πω απλά. Πρόκειται για μια έκθεση για την εγκαθάριση των λογαριασμών. Αυτό που λέμε ξεκάθαρα είναι ότι αυτή τη στιγμή μάλλον, σε καμιά φάση, στη διάρκεια 8 ετών, η Κομισιόν δεν λέει Ιδού το ποσό των γεωργικών δαπανών που αφιερώθηκαν σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της χρήσης ΤΑΔΕ. Αυτές οι οριστικές αποφάσεις όπου η Κομισιόν θα εκαθάρισε τους λογαριασμούς λέγοντας εμείς το 2007 δαπανήσαμε 54,8 δις ευρώ στον τομέα της γεωργίας. Αυτή η απόφαση δεν λαμβάνεται. Υπάρχουν διάφορες αποφάσεις που έχουν αποκλείσει παράτυπες δαπάνες, αλλά τελικά δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσό των δαπωνών που αναγνωρίζεται και αυτό δημιουργεί πρόβλημα επί το οποίο επέμεινε και η εισηγητριά σας. Ότι δηλαδή πουθενά η αρχή η αρμόδια για την απαλλαγή, δηλαδή εσείς και το Συμβούλιο, δεν μπορείτε να εκφραστείτε για ένα οριστικό ποσό. Αυτό είναι ένα σημείο που θεωρούμε ως σημαντικό, γιατί το απαιτεί εξάλλου και ο δημοσιονομικός κανονισμός, υποτυπικής τυπικής άποψης. Επίσης, θα ήθελα να επιμείνω για το γεγονός ότι οι διορθώσεις θα πρέπει να ορίζονται αντικειμενικά. Και το συνέδριο συμφωνεί απόλυτα με αυτό, αλλά διαπιστώνει πως σήμερα αυτή η αντικειμενικότητα δεν είναι σίγουρη. Και αυτή η αντικειμενικότητα δεν εξασφαλίζεται διότι είναι μια κρίση της Επιτροπής. Μια κρίση που εκφέρει η Κομισιόν για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των κρατών μελών. Εάν θεωρεί πως αυτή η αυτό το σύστημα ε, ελέγχου έχει αδυναμίες, τότε θα επιβάλλει μια αυθαίρετη διόρθωση και θα πει «Εκτιμώ ότι το ποσό των πιθανών ασφαλμάτων είναι 10%». Γιατί 10%? Εντάξει, τώρα υπερβάλλω κάπως, έχουν εμπειρία και έχουν ε, και βάσιμους λόγους για να πούνε ότι είναι 10% και όχι 20% και όχι 5%. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια κρίση, δεν βασίζεται σε κανένα αντικειμενικό κριτήριο. Και γι' αυτό και αυτό αμφισβητείται συχνά από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και όπως σας το είπα και πριν από λίγο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορες δικασίες δικαστικές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ορισμένα κράτη-μέλη αμφισβητούν τα ποσά διορθωτικά που τα επιβαρύνουν. Αυτό που συστήνει λοιπόν το συνέδριο είναι να περάσουμε από αυτές τις εκτιμήσεις σε κάτι πιο αντικειμενικό και για να έχουμε κάτι πιο αντικειμενικό πρέπει να εξετάσουμε τις, ε, τις συναλλαγές και να δούμε τις πραγματικές ε, διαδικασίες, τις πραγματικές συναλλαγές που έχουν γίνει και ποια είναι η πορεία των χρημάτων μέχρι το τελικό δικαιούχο της πληρωμής. Δεν λέει τώρα το συνέδριο πώς θα πρέπει να δουλέψει. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό ε, για την Κομισιόν, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ έχω διάφορες προτάσεις να κάνω. Εγώ εδώ να σας κάνω μία πρόταση. Πιστεύουμε, για παράδειγμα, πως μία δυνατότητα θα ήταν να αναθέσει στους εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης ένα ρόλο πολύ πιο διευρυμένο σε σχέση με αυτό που έχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό ο ρόλο ήδη έχει διευρυνθεί, το έχω υπογραμμίσει το 2007. Διευρύνθηκε ο ρόλος των οργανισμών πιστοποίησης και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να ζητήσουμε από τους εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης να εκφραστούν για την νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών των υπηρεσιών πληρωμής. Πράγμα που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Και έτσι η Κομισιόν θα έχει ένα ρόλο εποπτείας τις σωστές λειτουργίες αυτών των εργασιών που κάνουν οι οργανισμοί πιστοποίησης. Δηλαδή να εξασφαλίζει πως αυτές οι εργασίες βασίζονται σε δείγματα αντιπροσωπευτικά για τις διάφορες ε, ε, συναλλαγές και συνοδεύουν και θα συνοδεύεται και από ελέγχους επιτόπου. Έτσι ώστε να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν θα ξαναγράψω εγώ τον κανονισμό της κοινή γεωργική πολιτικής μετά το 2013. Αυτό είναι έργο της Κομισιόν. Εγώ περιορίζομαι να πω κάτι συγκεκριμένο. Για να σας πω κάτι συγκεκριμένο, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Αυτό θα κατέληγε στο να καθοριστεί πιο αντικειμενικά το ποσό των διορθώσεων. και επιτάει και η διαδικασία θα είναι πολύ πιο σύντομη γιατί έτσι θα εξαλειφθεί η φάση της συνδιαλλαγής όπου σήμερα αυτή η φάση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Κομισιόν εμείς την έχουμε αποκαλέσει μια φάση διαπραγμάτευσης ο κύριος ε, Μέγκλε διαμαρτυρήθηκε για αυτό το, φράση διαπραγμάτευση ωστόσο ισχύει σε κάποιο βαθμό, είναι διαπραγμάτευση Εξαρτάται ποιο έννοια δίνουμε στη λέξη συνδιαλλαγή. Ανάμεσα στο συνδιαλλαγή και στο διαπραγμάτευση υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Και αυτό ε, παρατείνει τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν θα συντόμευαν οι διαδικασίες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ χρονοβόρες. Σε αυτά είχα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ. Από τους βουλευτές υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο. Εγώ έχω μια ερώτηση να θέσω. Μια ερώτηση για τους οργανισμούς πιστοποίησης. Χάρη στην Ίγκε, επισκεφθήκαμε αυτή της Γαλλίας, δεν αν το θυμάσαι, αλλά στην έκθεση αγγίζουμε τα, τα θέματα ηθικής και ανεξαρτησίας. Ε... Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι οργανισμοί απέναντι στους εθνικούς κρατικούς μηχανισμούς ώστε να μπορέσουν να κάνουν σωστά τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουν και έπειτα στη σειρά στην αλυσίδα ελέγχου σε ποια φάση θα μπορούσαμε μέσα στο γενικότερο προβληματισμό μας να εμπλέξουμε τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Καταρχήν, η ανεξαρτησία των οργανισμών πιστοποίησης είναι μια απέτηση του κανονισμού. Ο γεωργικός κανονισμός προβλέπει ότι οι οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι από τις υπηρεσίες και από τις, ε, τους διοικητικούς μηχανισμούς που ελέγχουν. Εν γέννη αυτό συμβαίνει, ισχύει. Η Κομισιόν συχνά ε, παίρνει ερωτήσεις για αυτό το θέμα, αλλά δεν έχει ρόλο από λήψης απόφαση Δηλαδή δεν μπορεί να απορρίψει έναν οργανισμό πιστοποίησης με το αίτιο ότι δεν θεωρεί ότι είναι αρκετά ανεξάρτητος αλλά εξετάζει το θέμα και αν θεωρεί πως δεν είναι αρκετά ανεξάρτητος μπορεί να κάνει παρατηρήσεις κτλ. Πάντως δεν έχει δικαίωμα απόφασης. Αυτό το θέμα είναι θέμα των κρατών. Σε ορισμένε περιπτώσεις λοιπόν είδαμε ότι μπορούσε να υπάρξει κάποια βελτίωση στην ανεξαρτησία των οργανισμών πιστοποίησης. Α, και ο ρόλος των ελεγκτικών συνεδρίων. Είναι ένα πρόβλημα αρκετά περίπλοκο. Όπως το γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι εξαιρετικά υπέρ κάτι τέτοιο. Να σας πω γιατί. Διότι αυτό το σύστημα των εθνικών οργανισμών πιστοποίησης των, ελεργο... των ε, λογαριασμών των ε, ε, υπηρεσιών πληρωμών, ε, σε ποιον αναφέρονται στην Κομισιόν. Για μας, για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Κομισιόν. Και ο εξωτερικός ελεγκτής είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν είναι τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια θα μπορούσαν να συμμετέχουν, αλλά για να συμμετέχουν θα έπρεπε να υπάρχουν και να πληρούνται κάποιοι όροι, μεταξύ των οποίων είναι ότι τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια θα πρέπει να ανοίξουν τους φακέλους τους στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, να επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να πάει επί τόπου και να εξετάσει τη δουλειά που έχει γίνει, να εξασφαλίσει δηλαδή πώς είναι πλήρης η εργασία, αντιστοιχεί στους κανόνες που ισχύουν για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οπότε βλέπετε τι είδους διπλωματικά προβλήματα θα, θα δημιουργούνταν. Και για να μιλήσω και για ένα μόνο ελεγκτικό συνέδριο, αυτό το οποίο γνωρίζω πολύ καλά σε εθνικό επίπεδο, δεν ξέρω αν οι επόπτες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ήταν πολύ ε, ευπρόσδεκτοι αν έφταναν ε, χαροπά ε, στο Παρίσι. Και φαντάζομαι το ίδιο θα συνέβαινε και αλλού, όχι μόνο στο Παρίσι, όχι μόνο στη χώρα μου. Η παρέμβαση λοιπόν των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων θα δημιουργούσε μέγα πρόβλημα διότι υπάρχει πρόβλημα ιεράρχησης ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Εθνικά. Μέχρι στιγμής λοιπόν κρατάμε ε, δεν είμαστε ευνοϊκοί για αυτή τη λύση. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Φυσικά, ναι, εμείς συμβουλεύουμε βουλευτέ ε, έχουμε κάτι να πούμε πάνω σε αυτά. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Κομισιόν τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο μα μίλησε. Πήραμε και αυτή τη δήλωση προ τον τύπο τη Κομισιόν, η οποία απαριθμεί με ακρίβεια ποια κράτη μέλη έχουν καθυστερήσει για ποια ποσά ή πόσα, ποια ποσά του ζητιούνται να επιστρέψουν. Η ερώτησή μου είναι ποια είναι τα χρονικά όρια με τα οποία ζητάτε η ανάκτηση των ποσών αυτών. Λέτε ότι ζητάτε εδώ 214 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε ποια χρονικά όρια τα ζητάτε αυτά τα χρήματα και πώς μπορείτε να περιγράψετε με ακρίβεια αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απάντηση είναι απλή. Τρεις μήνες μετά την απόφαση. Και αυτό που γίνεται είναι ότι οι μηνύες πληρωμές προς τα κράτη-μέλη περικόπτονται ε, βάσει του ποσού αυτού που διερθώνεται. Είναι δηλαδή ένα θέμα λογιστικής. Έτσι κατακρατούμε δηλαδή, αυτά τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσουμε στα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνετε την ισχύ της Κομισιόν. Oui, monsieur Άρα είναι μια ιδανική κατάσταση αυτό και στρέφουμε εδώ προς τον κύριο Τεβέρ. αν γινόταν αυτό και σε άλλους τομείς, ε, θα ήταν θαυμάσιο, παραδείγματος στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Η πρακτική αυτή όμως είναι μεταφέρσιμη και σε άλλους τομείς. Στον τομέα της ε, γεωργίας τουλάχιστον ακολουθούνται κάποιες άουξες που μας φαίνονται απόλυτα λογικές και θα θέλαμε να σας αντέγραφαν και άλλες γενικές διευθύνσει οι οποίε δεν το κάνουν αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να δράσετε κύριε Είναι λεπτό πάντα το θέμα κύριε Πρόεδρε. Όταν ε, ε συγκρίνονται διαφορετικές δραστηριότητε που βασίζονται σε διαφορετικές ανάγκες και γι' αυτό για το 2013 η Κομισιόν έχει προσανατολιστεί για τον προπολισμό σε κάποιες από τις γραμμές ε, της, ε, ΚΑΠ, ε, της πολιτικής ΚΑΠ. Για πρώτη φορά, παραδείγματος χάρη, η Κομισιόν προτείνει στη βασική νομοθεσία, στην οριζόντια δηλαδή οδηγία που θα εφαρμοστεί για όλα τα διαφορετικά ταμεία, μια καθαρή διόρκωση θα μπορεί να γίνει εάν κάποιες τεσταλίδες έχουν επιπτώσεις στους τίσιους λογαριασμούς. και αυτή θα μειώσει τις δαπάνες στα ε, εν λόγω κράτη-μέλη. Ενώ τώρα επιτρέπεται να αντικατασταθεί αυτή η ε, μη κανονική δαπάνη, αν θέλετε, με άλλες δαπάνες. Ε, στην πρώτη της Κομισιόν δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει μια κύρωση. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια πρόταση Κομισιόν. Και από εκεί πέρα βέβαια ο νομοθέτης θα πρέπει να εκφράσει την άποψή του κατά πώς θα πρέπει να μεταφραθεί, μεταφραστεί συγγνώμη, σε νομοθετική πράξη όχι. Βέβαια αυτό δεν είναι τώρα η συζήτηση σήμερα. Το θέμα είναι πάρα πολύ πολύ πολύπλοκο και είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε από την εργασία σας ως συγγητής την περασμένο χρόνο πόσο πολύ είναι το θέμα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, μία σύντομη ανέθεση πάνω στο θέμα της ανεξαρτησίας που με ενδιαφέρει. Εγώ δεν αναφέρθηκα στην ανεξαρτησία των οργάνων πιστοποίηση σχετικά με την Κομισιόν, αλλά σχετικά με την διοικητική ιεραρχία των χωρών. Και όταν βλέπουμε το κράτο μέλο στο οποίο ανήκω εγώ, οι υπάλληλοι των αρχών πιστοποίηση ήταν οι υπάλληλοι που είχαν οριστεί από την ιεραρχία του και βέβαια υπό την επίδραση του Υπουργού. Τέλο πάντων, καταλαβαίνετε, αυτό είναι που με ενδιαφέρει και ιδίω όσον αφορά τους ε, όρους και τη διάρκεια ε, πληρωμών. Θα πρέπει δηλαδή να ελέγχει κανένα ότι τα όργανα αυτά είναι απόλυτα ανεξάρτητα. Μέσα δηλαδή στο ίδιο το κράτος μέλος σε σχέση με την εθνική ιεραρχία. Παρακαλώ με δύο λόγια. Έχετε δίκιο. Στη Γαλλία, Φερρυπίν, πρόκειται για υπαλλήλου του Υπουργείου ε, Γεωργίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά κυρίως ε, τους, ε, του σώματος ελέγχου. Αρκετά υψηλά ιστάμενοι ε, υπάλληλοι, δηλαδή που έχουν κάποια θεωρητική ανεξαρτησία σε σχέση με τον υπουργό τους και δεν εξαρτάται ο μισθός τους ανάλογα με το πόσο σαν σφάλματα θα βρουν. Όχι. Έχουν τον ίδιο μισθό σαν να έκαναν ό,τι κάνουν καθημερινά. Υπάρχουν δηλαδή πολλέ δυνατότητε για ανεξαρτησία, αλλά έχετε δίκιο, είναι κρατικοί υπάλληλοι, η οποία τελευταία ανάλυση εξαρτώνται από τον εκάστοτε υπουργό. Σωστό. Και βρήκαμε κάποιες παρόμοιες καταστάσεις σε μία σειρά κρατών μελών. Μέχρι στιγμής, από όσο ξέρω, η Κομισιόν δεν αμφισβήτησε το ότι οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας των οργανισμών αυτών πιστοποίησης ήταν επαρκές και Γκρέσλε. Να ολοκληρώσετε. Όχι. Αυτό το θέμα της ανεξαρτησίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι υπηρεσίες αυτές της επιστοποίησης συνεδριάζουν συχνά και με κάλεσαν κάποιες τις φορές και λένε ξεκάθαρα ότι και λόγω της αρχής τους αισθάνονται πολύ πίεση όταν βρούνε κάτι. Και αν σε κάποιο κράτος γίνονται καθ... συχνά τέτοιου είδους διορθώσεις, μου λένε αυτός ήταν πέρσι, τώρα δεν είναι πια εκεί γιατί ε, πήρε μετάθεση προς τα έξω και θα πρέπει εμείς να τους προστατεύσουμε και γι' αυτό έχουμε ε, μία πρόταση στον κανονισμό για τον προβλησμό μας όπου λέμε θέλουμε να ξέρουμε ποιος αλλάζει και γιατί. Τι άλλη δυνατότητα έχουμε. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος ήταν και τώρα δεν υπάρχει πια. Αυτό που θέλουμε, δεν τολμώ να το πω, είναι να έχουμε εκεί υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν ο πιο αποτελεσματικό τρόπο για να οργανωθούμε. Γιατί όπω έχει σημαίνει η κατάσταση δεν μπορούμε νομίζω να πετύχουμε και μεγάλη πρόοδο. Τώρα δεν ξέρω πώ θα οργανωθούμε καλύτερα. Και άμα δω ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε ήδη τώρα για να επιβληθούμε. Χαίρομαι για το υπόλοιπο της συζήτησης. Και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε κάτι που είπε ο κ. Μέργη στην αρχή, με, σχετικά με τον έλεγχο 100% εξάντερ. Ναι, θα με είχε εντυπωσιάσει αυτό αν είχα εξαιρεθεί με το θέμα μόνο ένα χρόνο τώρα. Αλλά δυστυχώς αυτό το παράδειγμα 7 που εξέτασε ήταν να συγκρίνει τα αποτελέσματα της εξάντερ 100% με τους ελέγχους που γίνονται προηγουμένως και ε, πολλά θα μπορούσε να πει κανένα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαστε ε, απόλυτα περήφανος για το 100% ελέγχων εξ άντε. Θα πρέπει νομίζω να καταργηθεί γιατί τα αποτελέσματα δεν αναλογούν στις προσπάθειες. Και ε, για σχετικά με το πώς γίνονται επιτόπου, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει γιατί εκεί βρίσκονται τα σφάλματα. Γιατί βλέπουμε ότι η έλεγχη επί χάρτου, τι να σας πω, δεν είναι ίσως επαρκή. Ίσως κάτι να μας πείτε σχετικά. Λέτε 50% μετά από τόσα χρόνια. Αλλά κάθε χρόνο πόσες είναι οι διαφορές που υπάρχουν στους ελέγχους επιφανειών και ποσών. Γιατί τι λέμε, θα έχουμε ένα καινούριο κανονισμό, αυτό που έχουμε δει δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον παλιό κανονισμό, αλλά έχουμε πολλές ευκαιρίες για τον καινούριο κανονισμό και αυτό λυπήθηκα ε, η έκθεση αυτή που αναφέρει πολλά συγκεκριμένα και αρχής θέματα δεν την είχαμε και νωρίτερα. Και ξαναλέω, δεν κατηγορώ εδώ το ηλεκτρικό συνέδριο. Ε, τώρα θα ήθελα να σας πω όσον αφορά τον ε, κανόνα των 24 μηνών και όχι, γιατί όχι 36 μήνες. Η προστασία θα ήταν μεγαλύτερη με 36 μήνες. Ε, θυμάμαι, υπήρχε συζήτηση, η Κομισιόν πρότεινε 36, το Συμβούλιο κατέληξε στα 24. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να έχουμε 36 και 48 μήνες και όχι 24 γιατί και εδώ μπορεί κανένας να κρίνει ποιες, τι διακυβεύεται οικονομικά. Ε, φοβούμαι ότι ίσως δεν δίνονται επαρκή στοιχεία. Το σύστημα καλό είναι, θα ήταν ίσως καλό να το βελτιώσουμε. Δεν θα κανώ να εφαρμόσουμε κάποια από τα μέτρα. Και να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το εθνικό επίπεδο και τι διακυβεύεται εκάστοτε. Αυτό θα μας έδινε νομίζω καλύτερες δυνατότητες παρέμβασης. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση γιατί είναι βασική σημασία σε έκθεση το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πια τίποτα με τον παλιό κανονισμό και δεν γνωρίζουμε το καινούριο. Και έτσι θα ξαναβρεθούμε εδώ σε 5-6 χρόνια και θα συζητάμε τα ίδια θέματα και τα ίδια στοιχεία και δεν θα έχουμε ακόμα προχωρήσει περισσότερο φοβούμε. Και το πρόβλημα είναι ότι θα δούμε ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μικρή πρόοδος. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ίγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτό που είπατε, κυρία Γκρέσλα, πριν από λίγο. Στου ελέγχου εξάντα θα πρέπει να κάνουμε την εξή διάκριση, γιατί εξαρτάται από το σύστημα ελέγχου. Στου ε, επιφανειακού ε, ελέγχου, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, μπορούμε να πούμε ότι η διοικητική έλεγχη βάση είναι εξαιρετικά έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη φυσικά η ενημέρωση των κτηματολογίων και η καλή λειτουργία τους. Εκεί υπάρχει προστιθέμενη αξία σε άλλους ε, κανόνες, ωστόσο δεν έχει τόσο νόημα για τους 24 μήνες. Έχετε δίκιο. Είχαμε προτείνει 36 μήνες, το Συμβούλιο τους είχε μειώσει σε 24 στην παρούσα φάση. Κοιτώντας την γενικότερη εικόνα, δεν είδαμε ε, να υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, να περάσει η λύση των 36 μηνών και αποφασίσαμε την ενέργεια αυτή να τη σπαταλήσουμε, να την δαμπανίσουμε, αν θέλετε, σε άλλους τομείς. Στον καινούργιο κανονισμό που προτείναμε, Είμαι λιγότερο απεσιόδοξο από ότι εσεί, κυρία Γκρέσλα, γιατί στο άρθρο 9 βρίσκεται ακριβώς αυτό που αναφέρατε, ότι στο μέλλον οι αρχές πιστοποίηση θα τοποθετηθούν για την νομιμότητα και την τυπικότητα των συναλλαγών, συναλλαγών που διεξήχθησαν. Άρα ο στόχος είναι ακριβώς αυτός, το είπα και εξ αρχής, να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου οι αρχές πιστοποίησης θα εξετάζουν εντελεχώς το τι έκαναν ε, οι ε, αρχές και θα μας δίνουν ένα ποσοστό σφάλματος το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε μετά για τη διόρθωση. Αυτό είναι ο απότερος στόχος και μετά θα ακολουθήσει μια κατάταξη όπου καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγχει τις ε, ε, αρχές πιστοποίησης και οι αρχές πιστοποίησης τις αρχές που καταβάλουν τις πληρωμές και αυτές με τη σειρά τους τους ε, αγρότες. Άλλο ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Είπατε ότι οι διορθώσεις δεν είναι αντικειμενικές. Φυσικά μπορούμε να τσακωθούμε για το τι σημαίνει αντικειμενικός. Αλλά θεωρώ ότι είναι αντικειμενικές γιατί βασίζονται σε ένα λεπτομερές έγγραφο εργασίας όπου παρουσιάζεται με ακρίβεια ποιες περιπτώσεις ε, υπόκεινται σε ποιο, ε, σε πιο επίπεδο ποσοστού. Αυτό εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, το έχει δεχτεί και το δικαστήριο. Φυσικά δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη γιατί χάνουν χρήματα. Ασφαλώς. Και γι' αυτό ε, πηγαίνουν στο δικαστήριο. Και επίσης να ξέρουμε όταν παλιότερα ε, ε, όταν παλιότερα ελέγχαμε όχι με βάση το σύστημα αυτό, αλλά με βάση το με μονομένους ελέγχους και πάλι υπήρχαν πρόσφυγες στο δικαστήριο σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 για τη διάρκεια των ελέγχων. Το ελπίζω αυτό. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Αλλά βλέπω ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που μας ε, συστήνει πιο έντονο έλεγχο των αρχών πιστοποίησης και αυτό θα ακολουθήσει, ε, θα έχει ως συνέπεια πιο πολλές διαδικασίες διατησίες και πιο πολύ χρόνο. Όλα αυτά, θα επαναλάβω, αποτελούν κινούμενο στόχο. Προσπαθούμε να κάνουμε ε, όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τις βελτιώσεις που ε, πρέπει να γίνουν, αλλά ο δρόμος προφανώς ομολογμένος είναι μακρύς. Υπάρχει η πρόταση αυτή επιτάπητος, η οποία συζητιέται όχι μόνο στο Συμβούλιο, αλλά στην κανονική νομοθετική διαδικασία, στην οποία το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και έτσι νομίζω ότι τα κράτη-μέλη ε, θα αναγκαστούν να υποστούν πιο πολλές πιέσεις. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο η συγκεκριά, μάλιστα δεν θέλει. Να κλείσω λοιπόν. Ευχαριστώ για την εξαιρετική έκθεση που αποτέλεσε αντικείμενο αυτή τη παθιασμένη συζήτηση. Σα ευχαριστώ και ολοκληρώνεται έτσι η εξέταση του σημείου 8 και διακόπτω με 30 δευτερόλεπτα για να δώσω την προεδρία στον πρόεδρο της Επιτροπής. Να ξαναξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Οντί που με αντικατέστησε γιατί Ήμουν σε κάποιες επίκουσες εργασίες στη Βόρεια Ολλανδία. Δεν μπόρεσα να έρθω πιο νωρίς και τώρα περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, η ειδική έκθεση υπαριθμών 8 σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των επιστροφών στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική. Φαντάζομαι ότι θα ήθελα να κάνει κάποια αρχικά σχόλια η Ingeborg, αλλά να δώσουμε το λόγο πρώτα στο ελεγκτικό συνέδριο. Ποιο είναι υπεύθυνο, έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Θα παρουσιάσω την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τις ανακτήσεις ε, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Τρεις αρχές εξετάζει η έκθεση καταρχάς πόσο αποτελεσματικά είναι τα σύστημα τα οποία εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για την ανάκτηση των οφειλών. Κατά δεύτερον, πόσο επιτυχή είναι τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των ε, ε, πληρωμών και κατά πόσο ε, αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά με σωστό τρόπο. Κατά τρίτον, πόσο αποτελεσματική είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιτήρηση και την υποπτία της διαδικασίας αυτής. Εισαγωγικά θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί από το 2004, οπότε και έγινε ένας παρόμοιος έλεγχος τότε. Δεν υπήρχε δομή στους ελέγχους και οι πληροφορίες που δημοσιεύονταν δεν βασίζονταν σε βάση δεδομένων ενημερωμένες και ορθές. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται από το 2006 και μετά εισήγαγε τον κανόνα του 50-50. Μετά από τέσσερα χρόνια σε κανονικές συνθήκες ή μετά από 8 χρόνια όπου υπάρχει ε, δικαστική υπόθεση, τα κράτη-μέλη χρειάνονται 50% του ποσού. Αυτό προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιε αδυναμίες και κάποιοι κίνδυνοι ε, εγγενεί που θα πρέπει να προσέξουμε. Το τρίτο ζήτημα τώρα, το χρέος που προκύπτει από παρατυπίες και σφάλματα. Το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι κατά μεγάλο βαθμό τα κράτη-μέλη πληρούν και τηρούν τους κανονισμούς. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ διαφορετική η ερμηνεία των κανόνων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη ημερομηνία ε, ε, καταγραφής του χρέους ε, στους διαφόρους λογαριασμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση μειώνει την δυνατότητα την πιθανότητα επιτυχούς ανάκτησης και την εφαρμογή του κανόνα 50-50 για το δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρεται στο κατά πόσο είναι επιτυχή τα κρατη για να ανακτήσουν τις, ε, τα κατεβληθέντα ποσά. Είναι αρκετά χαμηλό το ποσοστό αυτό, μόνο 10%. Ωστόσο, από την εισαγωγή του νέου συστήματος το 2006 και μετά, τα ποσοστά ανάκτησης έχουν αυξηθεί και τώρα ανέρχονται σε άνω του 40%. Όπως και να έχει, όπως σωστά υποδεικνύει και στο έγγραφο εργασία η ακόμα και με το νέο σύστημα και με τους καλύτερα ποσοστά ανάκτησης της, τα κράτη-μέλη και οι δικαιούχοι μάλλον κρατάνε παραπάνω από το 50% των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ανάκτησης και την ε, διαγραφή, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι κανόνες δεν ήταν αρκετά ρητοί και έτσι το ελεκτικό συνέδριο κατάληξε ότι από το 2005 έως το 2009 ε, ε, πάνω από 100 εκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια ευρώ διαγράφονταν ετησίω. Και αυτό επιβαρύνει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι διαγραφές αυτές ε, ήταν μη αιτιολογημένες ή αποτελούσαν αποτέλεσμα αμέλειας. Εγώ θα ήθελα να είμαι σαφή στο σημείο αυτό ότι δεν θέλουμε να επέμβουμε στις εθνικές νομικές διαδικασίες, αλλά κατά τη γνώμη μας το κράτος ε, όπου συμβαίνει η παρτιπία, μάλλον το σύστημα ε, ελέγχου των παρτιπιών θα πρέπει να είναι πιο εναρμονισμένο. Και το ελεκτικό συνέδριο εξέτασε τις ε, ευθύνες και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, εποπτεία και την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάκτησης. Και ένα από τα πορίσματα ήταν ότι πάνω από το 90% των ποσών, τα οποία στο παρελθόν παρουσιάζονταν στους ετήσιους λογαριασμούς υπό τις ανακτήσεις, ήταν τελικά διορθώσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι διορθώσεις αυτές επιβαρύνουν τον φορολογούμενο και όχι από αυτόν που ε, είναι υπεύθυνο για την ε, παράτυπη καταβολή. Αυτό έχει βελτιωθεί από το 2009 και μετά, αλλά ακόμα δεν ήταν δυνατόν να οριστούν τα ακριβή ποσά ανάκτησης. Ένα άλλο πόρισμα ήταν ότι τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στη λογιστική έκθεση ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτά που καταγράφονται στα κράτη-μέλη για τους λογαριασμούς αυτούς και αυτό για διάφορους λόγους και η συμφιλίωση, αν θέλετε, η ομογενειοποίηση αυτών των δύο ε, ε, ομάδων είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Το ελεγκτικό συνέδριο, κύριε Πρόεδρε, έχει προβεί σε διάφορες συστάσεις ε, για να βελτιωθεί η διαδικασία ανάκτησης. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητά από τα κράτη-μέλη να αναφέρουν, να κοινοποιούν τις ατασταλίες, τις παρατυπίες μόλις ε, εντοπίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, το ελεγκτικό συνέδριο προτείνει να υπάρχει ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα και προθεσμία για την αναφορά τέτοιων παρατυπιών και για την ε, κοινοποίηση της ε, ανάκτησης. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε τις συστάσεις αυτές στην νομική της πρόταση για την μελλοντική ΚΑΠ. Θα ήθελα να θέσω κι άλλο ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τις νέες νομοθεσίες που, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από έξι εβδομάδες. Θα ήθελα να εισάγει ένα σύστημα όπου ο κανόνας 50-50 θα καταστεί κανόνας 100%. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μετά από 4 χρόνια σε ψυχολογικές περιπτώσεις ή σε, μετά από 8 χρόνια σε περίπτωση ε, δικαστικής υπόθεσης, δικαστικής αγωγής, το κράτος μέλος θα χρεωθεί το 100% του ποσού που δεν έχει ανακτηθεί. Αυτό ακούγεται σωστό, αλλά να προσέξουμε, γιατί αν τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι θα χρεωθούν όλο το μη ανακτημένο ποσό, υπάρχει κίνδυνος να γίνει λιγότερη έλεγχη εξ αρχής. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί με τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Και είδαμε ότι με τον κανόνα 50-50 υπάρχει ένας κίνδυνος στα κράτη-μέλη να διαχειριστούν την, τα ζητήματα αυτά προς όφελό τους. Θα ήθελα πρώτα να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σας, να ευχαριστήσω και την κυρία Γκρέισλε, η οποία στο ρόλο της ως εισηγήτρια και πάλι προσέφερε και συνέβαλε προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την οποία τόσο και επενέσατε. Έχετε λόγο, κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω, ελεγκτικό συνέδριο, για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση, γιατί το βέλτιστο αποτέλεσμα το πετυχαίνουμε. Αν συνδυάσουμε τις δύο εκθέσεις για τις ανακτήσεις ε, και την προηγούμενη εκθέση, τότε μόνο έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Στις συστάσεις μου λοιπόν στο σημείο 1 μιλάμε για καλύτερα αριθμιστικά στοιχεία. Τι εννοούμε. Μετά από μακρά μια διαπραγμάτευση μετά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήμουν για το τι ποσοστό τελικά παραμένει στα χέρια του παραλήπτη. Αποφάσισα να γίνω, αν θέλετε, διατητής και συμπεριέλαβα και τα δύο αριθμητικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μόνο 40% των κατά καταβληθέντων ποσών παραμένουν παρά την στα και την παραλήπτη, ενώ το ελληνικό συνέδριο μιλά για 10%. Εγώ απλά αυτό που αναφέρω είναι ότι ακόμα και αν λάβουμε ως βάση τα καλύτερα αριθμητικά στοιχεία, το 40% δηλαδή, εξακολουθεί να υπάρχει ένα 60% για τα κατά καταβληθέντων ποσών. Μεταξύ 60 και 90% είναι το ποσοστό αυτό. Αλλά το καλό είναι ότι αν ε, λαμβάνει κανένας αχρέωστητος καταβληθέντων ποσών μπορεί να κρατήσει και συνήθως δεν τον ανακαλύπτουν και αν τον ανακαλύψουν δεν τον τιμωρούν. Ε, τρεις καλές ειδήσει δηλαδή για κάποια τμήματα της Ευρώπης. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό και αυτό έχει να κάνει και με τη διαδικασία και τη συζήτηση που έγινε για την ΟΛΑΦ. Είναι ενδιαφέρον το κεφάλαιο και είναι και σημαντικό κεφάλαιο. Εδώ και καιρό κάνουμε διάφορες και πολύ μεγάλες συζητήσεις για τέτοια θέματα ανάκτησης. Έχουμε πετύχει διάφορα αποτελέσματα στον αγροτικό τομέα δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε κάτι σημαντικά επειδή το αγροτικό σύστημα είναι όπως είναι. Αλλά για να αναγνωρίσουμε πόσο ενδιαφέρουσε είναι οι προτάσεις που γίνονται τώρα για το πώς μπορούμε να μάθουμε πιο πολλά για τα ποσά αυτά, τα καταβληθέντα ποσά και σε ό,τι αφορά τον κανόνα το 50-50. Εγώ προσωπικά απογοητεύτηκα από τα έργα της ε, Task Force γιατί παρακολουθώ τα, την εργασία της εδώ και πολλά χρόνια και ασχολούμαι με τέτοια θέματα ανακτήσεων. Έπαιξε σημαντικό ρόλο η Task Force και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με το ελεκτικό συνέδριο. Βλέπουμε ότι η νομοθεσία αυτή δεν είναι ενιαία, δεν είναι εναρμονισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το σημείο μια κριτική διάθεση. Κατά πόσο πετύχαμε πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι το θέμα αυτό των αχρεωστήτων και των βοηθέντων ποσών παραμένει για μας ένα πολύ βασικό σημείο. Αναφέρεται αρνητικά και η Ιταλία στο σημείο 7 ως κράτος ε, ιδρυτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. από όλου που ωφελούνται από το σύστημα των κανόνων του 50-50, η Ιταλία είναι η πρώτη. Άρα ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει συγκεκριμένα σχέδια για την Ιταλία. Ενδιαφέρουσα έκθεση, τη συστήνω ανεπιφύλακτα και σε αυτό το σημείο θα κλείσω, Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσει Η εκπρόσωπος είναι η κυρία Πατρίσια Μπουνιό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μπορούσα να είμαι σύντομη γιατί πιστεύω πως οι ανταλλαγές απόψεων μέχρι στιγμή ήταν πολύ σαφείς και οι εκθέσεις είναι εύγλωτες. Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε για αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα, εκτός από την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την εκαθάριση. Όπως είπε ο κύριος ε, Αλανίσιλα, η έκθεση της, ε, του συνεδρίου αφορά το σύστημα ανάκτησης που γίνεται από τα κράτη-μέλη προς τους ε, τελικούς δικαιούχους, τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν ε, συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για την καταγραφή, την ανάκτηση και την ε, ανάκτηση των χρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, καθώς και τον τρόπο έκθεσης, σύνταξη έκθεσης Κομισιόν για αυτά τα θέματα. Και τρίτη πτυχή είναι ο τρόπος με τον οποίο η Κομισιόν παρουσιάζει στους ετήσιους λογαριασμούς της τα στοιχεία σε σχέση με την ανάκτηση. Εν γέννη, το συνέδριο γνωρίζει ότι το σύστημα που έχουν φτιάξει τα κράτη-μέλη για να ανακτούν τα εντοπισμένα ποσά, καθώς και η διαδικασία της Κομισιόν έχουν βελτιωθεί από το 2006. Η συγγήτρια σας το αναγνωρίζει επίσης και ενθαρρυνόμεθα από αυτά τα αποτελέσματα και από αυτή τη διαπίστωση. Μάλιστα η Κομισιόν έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και πάντα είναι θετικό το να διαπιστώνουμε πως ε, απέφερε καρπούς. Ωστόσο, η Κομισιόν γνωρίζει και συμμερίζεται πολλές από τις διαπιστώσεις που έγιναν για το γεγονός ότι η κατάσταση δεν είναι τέλεια και ότι είναι δυνατόν να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Είμαστε δε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημά μας και θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει από δύο οπτικέ γωνίε. Καταρχήν, όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση, που είναι φυσικά πρωταρχικό συμφέρον μα, και δεύτερον, όσον αφορά την ανάκτηση από του δικαιούχου. Και γι' αυτό και σημειώνουμε με προσοχή τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και αυτές της κυρίας Γκρέσλε. Θα έλεγα ότι κατά βάση και χωρίς βεβαίω να, να ε, μην, να, μην, να προκαταβάλουμε το τελικό αποτέλεσμα της έκθεσης, ε, θα έλεγα ότι συμφωνώ με τις συστάσεις ε, του κυρίου Νίσηλα και έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις και φυσικά στο όρια των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν και της Γενικής Οικονομίας του Συστήματος ε, κοινή Διαχείρισης και Καθάρισης των Γεωργικών Δαπανών. Ποια είναι αυτά τα όρια και αυτές οι αποχρώσεις. Νομίζω πως είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε και τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και μέσα σε ποιο πλαίσιο. Πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι το να γνωρίζουμε και να δεχτούμε πως θα πρέπει να γίνει μια διάκριση και πιστεύω εδώ όλοι θεωρούν ότι το γνωρίζουν, αλλά είναι χρήσιμο να το θυμίσουμε, είναι ότι από τη μια πλευρά έχουμε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωση, για την οποία είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι ως Κομισιόν και έχουμε και περιθώριο λιγμών, αλλά και την πραγματική ανάκτηση από την άλλη πλευρά από τους δικαιούχους των τους καταβληθέντων ποσών, όπου αυτό εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία και στο εθνικό δικαστικό σύστημα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν δεν είναι αρμόδια, δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρέμβει στο εθνικό δίκαιο και δεν το επιθυμεί κιόλας. Δεν έχουμε, α πούμε, αρμοδιότητα για να παρέμβουμε στις εθνικές διατάξεις όσον αφορά την πτώχευση, που είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία που έχει θίξει το ελεγκτικό συνέδριο. Μέσα στο νομικό πλαίσιο αυτό είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε την πλαισίωση που μπορούμε να δώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή τα κράτη-μέλη ενεργούν και για να το οθήσουμε να ακολουθήσουν τον ορθό δρόμο. Όσον αφορά λιγότερο τα νομικά όρια και περισσότερο τις ε, αποχρώσεις ερμηνείας, όπως έλεγα, Ακόμα και αν το σύστημα δεν είναι τέλειο και θα ήταν επιθυμητόν ε, και εφικτόν να υπάρξουν βελτιώσεις, η Κομισιόν έχει μια αντίληψη κάπως πιο ε, διαφορετική από αυτήν του του συνεδρίου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι κίνδυνοι. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτοί οι κίνδυνοι καλύπτονται καταλήλως είτε μέσω των ελέγχων που κάνουν τα όργανα πιστοποίησης, αν και πάντοτε υπάρχουν πιθανότητες να ρωτηθεί κανεί και να προβληματιστεί και να βελτιώσει. Είτε λοιπόν από τα όργανα πιστοποίησης μέσα στο πλαίσιο της ε, οικονομικής εκαθάρισης των λογαριασμών, δημοσιονομικής συγγνώμη, εκαθάρισης των λογαριασμών, είτε μέσω ελέγχων που κάνει η ίδια η Κομισιόν μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας εκαθάρισης προς συμμόρφωση. Και θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι από τη στιγμή που διαπιστώνεται κάποια δυναμία ή κάποιο λάθος, ο οικονομικός κίνδυνος καλύπτεται από την δημοσιονομική διόρθωση. Διαφορετική βέβαια από την ανάκτηση από τους δικαιούχους, αλλά τουλάχιστον εγγυόμαστε τα, οικονομικά, τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Όπως σας είπα λοιπόν, επιθυμούμε να βελτιώσουμε το σύστημα και είμαστε σε θέση να πούμε ότι και ο κύριος Άλαν Ίσαλα το, το παρατήρησε ότι οι κύριες συστάσεις που κάνει το συνέδριο και που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση της κυρίας Γκρέσλε έχουν υιοθετηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πρόταση κανονισμού, μάλλον οριζόντιου κανονισμού που παρουσιάσαμε για την περίοδο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2013 και ένα παράδειγμα δόθηκε, αλλά θα μπορούσα να σας δώσω και κάποιο άλλο. Έχουμε ας πούμε το θέμα τη στιγμή όπου τα χρέη θα πρέπει να καταγραφούν, να κοινοποιηθούν στον δικαιούχο και να αναφερθούν στην Κομισιόν, που είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι έτσι ξεκινά όλη η διαδικασία ανάκτησης και έμεσα προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προτείνουμε λοιπόν σε ένα νέο άρθρο 56 του οριζοντίου κανονισμού διατάξεις πολύ πιο ξεκάθαρες και συγκεκριμένες που θα επιτρέψουν να ξεκινά στο τέλος ενό έτους αυτή η υποχρέωση καταγραφής και που θέτει τέλος σε κάποιες αμφισημίες που μπορούν να υπήρχαν στην έννοια της υποστήριξης και του τρόπου εφαρμογής και ερμηνείας στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Άλαν Ισαλά επίσης σημείωσε ότι προτείνουμε να αντικατασταθεί ο κανόνας αποζημίωσης του 50% στο τέλος των 4 ετών, ίσως και 8 ετών, σε περίπτωση ε, διαδικασίας δικαστικής μέσω του κανόνα της ανάκτησης 100%. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε, να οθήσουμε τα κρατημέλη να επιταχύνουν την ανάκτηση από τα κάτι μελη Διότι τα κάτι μελη γνωρίζουν ότι μετά από τέσσερα χρόνια δεν έχουν κάνει, δεν έχουν προβεί στην ανάκτηση, θα τους ζητηθεί η κάλυψη του 100% του χρέους. Είναι ένα κίνητρο σημαντικό. Δεν παραμαλούμε το γεγονός ότι Ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο ίσως σε επίπεδο 100 μελών το να προσπαθήσουν να κρύψουν περισσότερο ή να ε, παραλείψουν τον καταγραφή ορισμένων χρεών, αλλά αυτό το λαμβάνουμε υπόψη στις αναλύσεις κινδύνου μας και έτσι θα μπορέσουμε να επιτείνουμε τους ελέγχους για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν. Θεωρούμε, μετρώντας, ε, ζυγίζοντας ε, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους, ότι τα πλεονεκτήματα είναι περισσότερα από τα προβλήματα. Αυτά είναι δύο παραδείγματα που ήθελα να σας δώσω για τις βασικές αλλαγές, τροποποιήσεις που προτείνουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις ε, της, του συνεδρίου. Υπάρχουν και άλλες τροποποίησης. Οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν βεβαίως για όλες αυτές τις τροποποίησεις αλλά και για όλες συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των ε, ε, τόκων. Θα επανέλθουμε με κατευθυντήριες γραμμές που θα επιτρέψουν ε, την, να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν να κλείσω, και γενικά πιστεύω πως είμαστε σε θέση να πούμε πως είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και να λάβουμε υπόψη τις περισσότερες παρατηρήσεις που έγιναν όσον αφορά την Ιταλία που αναφέρθηκε από την κυρία Γκρέσλε. Δεν είμαστε αδιάφοροι για αυτό το πρόβλημα φυσικά. Ε, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Οι περιπτώσεις που παραμένουν, το γνωρίζετε βέβαια, είναι υποθέσεις που εμπίπτω στα όρια των όσων σας περιέγραψα εξ αρχής είναι θέματα που βρίσκονται σε δικαστική διαδικασία και ακολουθούν το ρυθμό τους ε, που είναι αργός πάντως ε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εξασφαλίζουμε ότι όλα αυτά γίνονται όπως πρέπει. Εν γέννη λοιπόν νομίζω πως είμαστε στο ίδιο μήκο σχήματος. Ε, θέλουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε στη διαδικασία ανάκτησης γιατί είναι αλήθεια ότι τα χρήματα αχρεωστήτως καταβληθέντα πρέπει να επιστραφούν. Ήδη στο πλαίσιο του προ... της πρότασης οριζόντιου κανονισμού έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και φυσικά και θα λάβουμε υπόψη κάθε επικοδομητική πρόταση και στο μέλλον. Εν τω μεταξύ όμως θα πρέπει να ξέρετε, γιατί όπως έλεγε και η κυρία Γκρέσλα, θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι ότου αυτές οι μεγάλες τροποποιήσεις να τεθούν σε εφαρμογή. Ωστόσο, μεταξύ, μέσα στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου προσπαθούμε να διορθώνουμε τις κατευθυντικές μας γραμμές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκρέσλε και κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα το λόγο έχουν τα μέλη που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Κύριος Γερμπράντη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ολυμπικό Συνέδριο και την Κομισιόν για την έκθεση και τις παρατηρήσεις. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κρέσλεν, την εισηγήτριά μας, για το σχέδιο έκθεσής της. Υποστηρίζω εντονά τις συστάσεις του συνεδρίου και της κυρίας Γκρέσλε. Έχω μία σοβαρή πολιτική ερώτηση. Γιατί οι παρουσιάσεις αυτών των θεμάτων πολλαπλασιάζονται και έχουμε συνεχώς το ίδιο πρόβλημα ότι τα κράτη-μέλη δεν φαίνεται ότι ενδιαφέρονται για τα ίδια πράγματα που ενδιαφερόμαστε εμείς. Και αυτό είναι να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα τα ευρωπαϊκά χρήματα και να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται μόνο να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα και όλα τα άλλα δεν του ενδιαφέρουν. Το ερώτημά μου είναι και προς το συνέδριο και προς την Κομισιόν είναι ότι ας πούμε μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα, να υποστηρίξουμε τις συστάσεις, να δυναμώσουμε το ρόλο της Κομισιόν δεν έχετε όμως την εντύπωση ότι εφόσον δεν συζητάμε το θέμα του διαστατικού προβλήματος, τη στάση δηλαδή των κρατών μελών, δεν έχει και μεγάλο νόημα να επιλύσουμε τις λεπτομέρειες. Δεύτερο ερώτημα. Είχατε κάποια αντίδραση από τα κράτη-μέλη όσον αφορά το ρόλο τους για το θέμα αυτό και αυτό το ερωτώ και προς το συνέδριο και προς την Κομισιόν. Και θα ήθελα να ρωτήσω, Πρόεδρε, εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, να προσπαθήσουμε να ξαναεπανέλθουμε στο θέμα. Ευχαριστώ. Πρώτα, εγώ σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να υποβάλει ερώτηση. Έχω εγώ μία ερώτηση που είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν κάποιο κράτος μέλος που το συνέδριο θεωρεί ότι έχει ένα νομικό σύστημα που θα πρέπει να ε, συστήνουμε σε άλλα Δεν μπορούμε να σε επιβάλλουμε βέβαια κάποιο σύστημα, αλλά μπορούμε να πούμε αυτό το σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Εμείς ε, εξετάζουμε την έκθεση του ηλεκτρικού Συνεδρίου εδώ στο Συμβούλιο. Αντέδρασε ποτέ όμως το Συμβούλιο για κάποια έκθεση του ηλεκτρικού Συνεδρίου πάνω στη θέματα αυτά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε ποια είναι η αποδεκτή στάση του Συμβουλίου. Του Συμβουλίου. Και θα πρέπει ίσως και το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει πάνω στα συμπεράσματα του συνεδρίου. Έχετε ακούσει κάτι. Ποια είναι η κατάσταση. Παρακαλώ. Ε, thank you, chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να συμφωνήσω με τα σχόλια που ακούσαμε. Ιδίω με αυτά που είπε η συγκέντρια, παρόλο που όλα βέβαια είπαμε δεν είναι ικανοποιητικά η Κομισιόν έχει προτείνει ένα χρονικό όριο μεταξύ της ανακάλυψης και της κοινοποίησης. Έχω κάποια προβλήματα, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα πολλά στοιχεία αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον είναι να δούμε την ε, κατάσταση στην οποία τα χρέη καταγράφονται το αργότερο δυνατό. Άλλα σχόλια αφορούν τον ρυθμό ανάκτησης, ε, ενώ την αργή, η ανάκτηση αυτή σε σχέση με τα ανοιχτά χρέη που πολλές φορές είναι πολύ παλιά. Προέρχονται από πριν από το 2006 Φερρυπίν. Αλλά βέβαια το 2006 ήταν γνωστό ότι τα ρυθμοί ανάκτηση ήταν 40 με 60%. Και τώρα υπάρχει ένα νέο σύστημα από το 2006. Τα τελευταία στοιχεία είναι του 2010 από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κομισιόν και έχουμε ένα ποσοστό 42% τα έτη 2007-2010. Υπάρχουν βέβαια πολλές δυνατότητες βελτίωσης. 42% δεν είναι ικανοποιητικό. Και αυτό οφείλεται ιδίω στι δυσκολίε τη εντολή. Γιατί βλέπουμε όχι μόνο οι παραγωγοί και οι εταιρείε και οι έμποροι προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν την ανάκτηση. Uh, uh, Τέλος, υπήρχε και δική σας ερώτηση, κύριε ε, Πρόεδρε και η ερώτηση του κυρίου Κρεπλάντη. Ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα με την Επιτροπή Γεωργίας, υπήρχαν καθυστερήσεις κλπ. Ε, η αντίδραση όμως ήταν καλή γιατί τα κρατημένα δεν αναγνώρισαν ότι χρειάζονται ε, μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ίσως πραγματικά θα μπορούσαμε να μάθουμε από τις ε, βέλτιστες πρακτικές. Ορισμένα κράτη-μέλη καταφέρουν να ανακτήσουν σχεδόν το 100%. Αυστρία, κατοχώρες, Φερρυπίν. Άλλες λιγότερο από το 20% ίσως πραγματικά υπάρχουν κάποιες βέλτιστες πρακτικές εκεί που μπορούν να τι υιοθετήσουν και άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ στα στοιχεία αυτά να προσθέσω ότι πράγματι η κατάσταση διαφέρει από κράτος σε κράτος. Η στάση ορισμένων μόνο είναι κάπως σχιζοφρενική. Δεν διαφέρονται για το θέμα το, δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια πόσο πολύπλοκοι είναι οι κανόνε ε, βάσει των οποίων κινούμεθα και που οδηγούν σε διαδικασίε ε, που σχετίζονται με αναγνώριση των χρεών, που πραγματικά μα κάνουν να κατανοήσουμε γιατί είναι τόσο πολύπλοκοι οι διαδικασίε. Ε, καμιά φορά ίσως δεν υπάρχει και η, η, η ιδιαίτερη ε, επιμέλεια. Βέβαια τα συστήματα δεν είναι 100% στεγανά, αλλά εξετάζουμε εμείς όλα αυτά τα στοιχεία που σας προανέφερα. Και λόγω του πολυπλόκου των κανόνων μπορεί να δοθεί κάποια εξείδηση για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ιδίω αυτά που αναφέρονται στη νέα μας πρόταση που προσπαθούμε κατά μέγιστο να απλουστεύσουμε τους κανόνες που εφαρμόζονται όσον αφορά την αναγνώριση του χρέους. Άλλα συστήματα, υπάρχουν συστήματα δικαίου για τα οποία ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τι μπορεί να γίνει. Τέλος, υπάρχει μία προσέγγιση απλούστευσης Τα συστήματα πληρωμής και υποστήριξης που ισχύουν αυτή τη στιγμή είναι απλά και εάν οι κανόνες ελέγχου είναι αποτελεσματικοί, τόσο πιο εύκολο μπορεί να βρεθεί σε κάποια λύση η προσέγγιση έχει πολλές πτυχές. Δεν εξαρτάται μόνο από την καλή θέληση ενός κράτους μέλους, παρόλο που και αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλέψουμε φυσικά. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορκ, δεν νομίζω θες να σχολιάσεις. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω το Ενεκτικό Συνέδριο, τον κύριο Αλανίσιο Λαϊδίος και την Κομισιόν και όλους και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα συνεδρίες εδώ και θα ζητήσω από τους συντονιστές να παραμείνουν για τις συνεδρίες των συντονιστών. Και όλοι οι άλλοι παρακαλώ μπορούν να φύγουν από την αίθουσα.